Good morning everybody. Guten Morgen. Kommen zur Tagesordnung des heutigen Tages. Καλημέρα. Είμαστε στην ημερήσια διάταξη σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως ξέρετε, υπήρξαν δυσκολίες όσον αφορά την έκθεση Κώστα. Είχαμε κάποιες προτάσεις από μία σκιώδησχηγήτρια, οι οποίες τελικά δεν μπόρεσαν να συζητηθούν. Γι' αυτό και θα αναβληθεί η πρωτοβουλία, η ψηφοφορία αυτή, συγγνώμη, και θα υπάρξει η αλλαγή αυτή θα την ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Καταρχήν όχι η έγκριση των πρακτικών, αν δεν υπάρχουν ε, με... Σήμερα έχουμε διερμηνία σε κάποιες γλώσσες, όχι σε όλες. Ολλανδικά μπορείτε να μιλήσετε, αλλά δεν υπάρχει ε, διερμηνία και δεν υπάρχει βεβαίως ακόμα στα κροατικά. Αν κοιτάξετε το φάκελό σας, θα βρείτε τις εκθέξεις, θα βρείτε την παρουσίαση της γραμματείας ε, για την αντιπροσωπεία στο Μάριμπορτ, πρέπει να σας ε, ενημερώσουμε καθότι όπως ξέρετε αυτά τα ταξίδια τώρα περνάνε από προηγούμενη συζήτηση και περιμένουμε την άδεια. Η κυρία Παλιαδέλη έχει την ε, πρώτη έκθεση. Θέλετε καταρχήν το λόγο πριν περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Όσον αφορά τα θέματα της ανθρωπιστικής ε, σε αυτό θα γίνει δεχτό. Λοιπόν, εντάξει, περνάμε τώρα στο θέμα της ψηφοφορίας. Όχι. Καταρχήν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ναι. Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά υπέρ επαναλαμβάνουμε υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος για το 16 Εντάξει, τέλος. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Μπάκο. Δεν πρόλαβε. Ωραία, ψηφίζουμε το 16 υπέρ. Κατά αποχές ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Υπέρ. κατά, εγκρίθηκε. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος για το 20. Τέλος. με τον κύριο Μπάγκο 17-9 εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 10 τέλος 13, 14 κατά Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ναι, σε μέτρησα. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 11. Τέλος. 13 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία τρια υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε το 3. Τέλος. 22-6. Κάτι λάθος έκανα. Ευχαριστώ. 13. Υπέρ. Κατά. Α, ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 13. Τέλος. 12 υπέρ 16 κατά. Απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά. Αποχές μία ψήφος κατά. Εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παλιαδέλη. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της κυρίας Παλιαδέλη και αυτό είναι στρατηγική καινοτομία πάλι για το Ινστιτούτο. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 37. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 20 το εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές α έλεγχος 45 ελέγχουμε ελέγχουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει η 3 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ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 Α, 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για το 56. Τέλος. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, τέλος. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Εγκρίνεται. 30. εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά. 2 κατά εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Παλιαδέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ist gar Και τώρα περνάμε στο σημείο 6, 7, 7, συγγνώμη. Έκθεση Φοντάνα. Θέλετε να μιλήσετε? Έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, κυρίως τη Στεφανή που μας βοήθησε όλους πολύ και όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο. <clears throat> Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 64. 47, 49, 50, 50 υπέρ. Απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τις, ε, την τις επόμενες από την 6 μέχρι την 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Έλεγχος για την 70. Τέλος. Απορρίπτεται η 70. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Για την 71. Τέλος.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 αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές Α, έλεγχος για την 79 ελέγχουμε τέλος απορρίπτεται προφορική 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 81. Τέλος. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τέλος. Εγκρίνεται 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές. 88. Ελέγχουμε την 88. Τέλος. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2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 κατά αποχές 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβεβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, απορρίπτεται. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε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 Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία του 8. Ενδιάμεση έκθεση του κυρίου Λόκεγκαρτ. Θέλεις να πεις κάτι, όχι δεν θέλεις. Ωραία, τέλεια. Περνάμε λοιπόν. Στην ψηφοφορία. 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά 23 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε τη 46. Τέλος. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 47 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 48 εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε, ελέγχουμε την 9. Τέλος. Εγκρίνεται η 9. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Δύο κατά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λόκεγκαρτ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα... Ο κύριος Μπέλετ δεν είναι εδώ. Αχ, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, είναι ο κύριος Λόκεγκαρ πάλι. Άλλη έκθεση Λόκεγκαρ. Πρόκειται για το γενικό προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία ψηφοφορία. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 4 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 6, 7, 8. Όχι, όχι. Δεν γίνεται όλες μαζί, ε. Δεν θέλετε να ψηφίσουμε όλες μαζί. 6 λοιπόν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές το 15 μπορούμε να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 11 υπέρ, 19 κατά, 12, 12, Έτσι κι αλλιώς απορρίπτεται. 16 υπέρ. Υπέρ. Α, έχει δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Α, εγώ είμαι. Λοιπόν, και τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι πιο συγκεκριμένη έτσι ώστε να αποφύγουμε παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Κύριε Κορέλ, μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα την πλήρη προσοχή σας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν σας παρακαλώ πολύ να με παρακολουθήσετε και αν είστε και πολύ ε, θαραλέοι μπορείτε να διαβάσετε και το κείμενο το οποίο σας έχω στείλει ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν το έχουμε τυπώσει. Λοιπόν, πρόκειται για το νέο πρόγραμμα της Επιτροπής για την κατάρτιση, τους νέους και τον αθλητισμό. Το Μάιο και τον Ιούλιο συζητήσαμε το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ εγώ βρέθηκα με τους σκιώδεις και πολύ εντατικά συζητήσαμε το θέμα. Αυτά τα οποία λοιπόν σας τα ε, παρουσιάζω σήμερα δεν είναι μόνο δικές μου ιδέες. Έχω συμπεριλάβει και τις ε, ιδέες των συναδέλφων και ελπίζω να το πέτυχα. Λοιπόν, καταρχήν προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 3 Οκτωβρίου. Για μας στη Γερμανία είναι μεγάλη γιορτή αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει υποβάλλετε παρόλα αυτά τις τροπολογίες σας. 6 Νοεμβρίου ψηφίζουμε. 6 Νοεμβρίου ψηφίζουμε χωρίς να έχουμε, όπως ξέρετε, τους τελικούς αριθμούς του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Το μόνο που θα έχουμε είναι κάποια ποσοστά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο σας έχω στείλει και το οποίο δείχνει με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Τώρα, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου θα μπορέσετε να μου στείλετε τροπολογίες. Και σκεφτείτε το εξής. Το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε είναι την πρόταση της Επιτροπής, όχι το δικό μου κείμενο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, περιοριστείτε στο απαραίτητο. Αυτά τα οποία εγώ έχω ενσωματώσει στο κείμενό μου, σκεφτείτε ότι ίσως συμπεριλαμβάνουν και κάποια από τα σημεία τα οποία θα θέλατε να υποβάλλετε. Όσον αφορά τη δομή του προγράμματος, η πρόταση της Επιτροπής για τους τρεις αυτούς τομείς, κατάρτιση, νεότητα και αθλητισμό, βάζει τρεις κατευθυντήριες ε, γραμμές, τρεις κατευθύνσεις, τις οποίες εγώ δεν θέλω να αλλάξω. Πρόκειται για την κινητικότητα στην κατάρτιση, την καινοτομία και την στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Για αυτά εμείς συμφωνούμε, τα υποστηρίζουμε. Στο εσωτερικό αυτών των κατευθυντήριων γραμμών υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που ενσωματώνονται μεταξύ κατάρτισης και νέων και εδώ βεβαίως μπαίνει και το πολύ αγαπητό κεφάλαιο ε, στον Τζομονέ, τον αθλητισμό. Πρέπει να σας πω ότι άμεσα με τον αθλητισμό δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δράση ή άρθρο στο πρόγραμμα της Επιτροπής παρόλο που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Εγώ λοιπόν ε, πρέπει να σας πω ότι κινητοποιήθηκα και πρόσθεσα ένα ολόκληρο κεφάλαιο ξεχωριστό για τον αθλητισμό. Όσον αφορά την γενική και επαγγελματική κατάρτιση και δεύτερον τον αθλητισμό και τους νέους. Γι' αυτό και αυτές οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές διατηρήθηκαν, όπως τις προτείνει Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχει γίνει συνδυασμό των διαφόρων μέτρων όσον αφορά παραδείγματο χάρη την επαγγελματική κατάρταση. Υπάρχει μια πολύ γενική προσέγγιση της Επιτροπής, πολύ ασαφής και καθόλου φιλική προς τον ε, ε, τελικό χρήστη. Εμείς λοιπόν, παρόλο που βεβαίως και υποστηρίζουμε αυτές τις τρεις κατευθυντήριες γραμμές, θέλουμε να τις συγκεκριμενοποιήσουμε. Υπάρχει βεβαίως εδώ μια πολύ μεγάλη πίεση ότι στο προσκήνιο όλης αυτής της προσπάθειας υπάρχουν οι ανώτατες σπουδές, η ανώτατη εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ε, παρουσίαση των διαφορετικών τομέων. Δεν θα αλλάξω τίποτα, επαναλαμβάνω, στις τρεις αυτές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θέλω να είναι πιο ορατό σε αυτόν που θέλει να διαλέξει το τι ακριβώς υπάρχει, πιο περιεχόμενο. Φυσικά και θα κρατήσουμε λοιπόν αυτές τις τρεις ε, κατευθυντήριες γραμμές θα διατηρήσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες, το Λεωνάρτο Νταβίντσι, το Εράσμος, το Κομένιος και τα προγράμματα που απευθύνονται στους ενήλικες και την διαβίου κατάρτιση. Οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με την εκπαίδευση γνωρίζουν στην Ευρώπη ένα πρόγραμμα, το Εράσμος. Το Κομένιους υπάρχει Υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα για τα άλλα προγράμματα, τα οποία δεν πρέπει να τα βυθίσουμε και να τα εξαφανίσουμε. Με το νέο άρθρο λοιπόν 5α, εγώ έχω ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτές τις άλλες ονομασίες και τα άλλα προγράμματα. Δεν αλλάζω τίποτα στην πολυπόθητη απλοποίηση. Στο άρθρο 5β οι συγκεκριμένοι στόχοι, τους οποίους θέλουμε να πετύχουμε στους διάφορους τομείς. Η Επιτροπή είχε προτείνει κάποιους αρχικούς στόχους που καλύπτουν βέβαια όλο το εύρος των προγραμμάτων και εγώ αυτό το κράτησα. Πρόκειται για άλλες γραμμές, κατευθύνσεις, προσανατολισμούς, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο στοχεύουν τους διάφορους τομείς. Για τις δραστηριότητες στο εσωτερικό των προγραμμάτων, η Επιτροπή προτείνει μια αρχιτεκτονική και εγώ την διατηρώ. Επαναλαμβάνω συνέχεια τα ίδια, ίσως επειδή ήμουν καθηγήτρια και ξέρω ότι η επανάληψη βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουν ε, οι μαθητές. Οι καθηγητρίες γραμμές λοιπόν θα παραμείνουν. Εγώ θέλω όμως να γίνουν ξεκάθαρες στον κάθε τομέα κατάρτισης ποιες είναι οι δραστηριότητες που υπάρχουν, που προτείνονται. Θέλω λίγο να μειώσουμε την ανώτατη εκπαίδευση και να υπάρξει η βασική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση σε πιο ισορροπημένη μορφή. Σκοπός μου είναι να είναι ορατή οι διάφοροι τομείς, οι διάφορες δραστηριότητες και να υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα και πραγματικά δεν παρουσιάζουμε εδώ έναν εξαντλητικό κατάλογο, δείχνουμε όμως σε όλο το εύρος του το πρόγραμμα και ποιες είναι οι δραστηριότητες που προτείνονται. Επαναλαμβάνω, θέλω να κάνω την πρόταση της Επιτροπής πιο φιλική προς τον χρήστη και να μην είναι τόσο ασαφής όλο. Επίσης, παρουσιάζουμε για το πρόγραμμα Εράσμους, επίσης οι ιδέες που προτείνονται εδώ είναι πολύ γενικές και πολύ καλές. Οι διάφορες εγγυήσεις, παραδείγματος χάρη για τη χρηματοδότηση, για όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό. Όλοι όμως ξέρουμε ότι το Εράσμους δεν απευθύνεται σε όλους. Το Εράσμους απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ως ένα βαθμό αυτές τις σπουδέ στο εξωτερικό. Με 200 ευρώ κανείς δεν μπορεί να ζήσει στο εξωτερικό. Άρα εδώ παρουσιάζονται οι δυνατότητες για φοιτητικά δάνεια, για χρηματοδότηση. Θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε βεβαίως πολύ σοβαρά με την Επιτροπή στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν αυτά. Ποιος θα δανείσει σε ποιον και ποιος θα μπορεί να πάρει δάνειο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πριν ψηφίσουμε θα πρέπει να συμφωνήσουμε τις ιδιαιτερότητες αυτού του προγράμματος. Σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Πάντως και νομίζω αυτό συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι. Τώρα περνάμε στους νέους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εδώ έχει δώσει αυτή την έμφαση η Επιτροπή, αλλά πραγματικά όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει το κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι διάφοροι στόχοι για τις τρεις αυτές κατευθυντήριες γραμμές. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη διατύπωση για τον κάθε στόχο, συγκεκριμένη περιγραφή του τι θέλουμε να πετύχουμε στον τομέα των νέων. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να απομακρυνθώ καθόλου από την απλοποίηση. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε στους πολίτες της Ευρώπης τι θέλουμε να πετύχουμε. Η πρώτη κατευθυντήρη γραμμή, η κινητικότητα στην μάθηση, οι ανταλλαγές νέων, εθελοντική εργασία. Αυτό είναι κάτι που εμείς το έχουμε προσθέσει και γι' αυτό και θέλουμε να κατονομαστούν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Συνεργασία για καινοτόμες διαδικασίες, συνεργασία νέων και η τρίτη κατευθυντήρια γραμμή είναι η στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Το Φόρουμ των Νέων και βεβαίως εδώ το θέμα της χρηματοδότησης κάποιων ε, φορέων και οργανώσεων δημόσιων. Εδώ αυτή η ιδέα προέρχεται από συναδέλφους. Οι οργανώσεις των νέων εδώ είναι κάτι που συμφωνήσαμε και με το Συμβούλιο. Πρέπει το πρόγραμμα αυτό να συμπεριλαμβάνει όλες τις δυνατότητες για τους νέους. Υπάρχουν και έξι φορείς εδώ, οργανισμοί που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα από το Jean το Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπρουζ, στη Φλωρεντία, στη Μάστριχτ, στην Τρίερ, η σχολή στη Δανία, στην Κοπενχάγη και η σχολή για την κατάρτιση στην Νίκαια. Πρόκειται εδώ για μια νέα πρόταση που προτείνει τη χρηματοδότηση μόνο των δύο πρώτων από αυτούς τους δύο οργανισμούς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως αυτές οι δύο είναι πιο δυναμικές και θα αντιδρούσαν πιο έντονα γιατί είναι πιο γνωστές. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι και για τους έξι αυτούς οργανισμούς, Ινστιτούτα, θα πρέπει να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτή την επιλογή. Και τώρα περνάω στον αθλητισμό. Η Επιτροπή είχε κάνει ένα πολύ μικρό κεφαλαιάκι για τον αθλητισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο αθλητισμός. Θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και εδώ θέλουμε να γίνει πολύ πιο σαφής η αναφορά στον αθλητισμό. Γι' αυτό και έχουμε ενσωματώσει δραστηριότητες, στόχους στον τομέα του αθλητισμού. Βλέπετε ότι για πρώτη φορά συμφωνούμε πιο πολύ με το Συμβούλιο παρά με την Επιτροπή. Οι δείκτες αυτών των στόχων, εντάξει υπάρχουν διάφορα τεχνικά αν θέλετε στοιχεία στα παραρτήματα, η πρόταση για τον αθλητισμό όμως θα πρέπει σαφώς να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ αθλητισμού και κατάρτισης, τον εθελοντικό αθλητισμό και θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες για όλους, εγκαταστάσεις και βεβαίως εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Γίνεται και μια ειδική αναφορά στους παραολυμπιακούς αθλητές. Τώρα βεβαίως εδώ, όπως σας είπα, η χρηματοδότηση, ή αριθμοί πρέπει να περιοριστούμε σε ποσοστά. Δεν έχουμε αριθμούς συγκεκριμένους και ο συνολικός προϋπολογισμός έχει κατανεμηθεί μεταξύ των νέων τις δραστηριότητες ζωμονέ, την κατάρτιση και τον αθλητισμό. Και υπάρχουν εδώ κάποια ποσοστά όσον αφορά την κατάρτιση, ο προϋπολογισμός έχει κάποια ελάχιστα ποσοστά ανατομέα. Στην Επιτροπή υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ελάχιστες ε, χρηματοδοτήσεις. Εδώ βλέπω 56%. Αυτό είναι το ποσοστό που προτείνει η Επιτροπή. Όμως δεν αναφέρεται παντού αυτό το ποσοστό. Η συμμετοχή, αν θέλετε εδώ, δεν είναι δεσμευτική. Η ανακοίνωση αυτών των ποσοστών για μένα πρέπει να γίνει εδώ έτσι ώστε να γίνει δεσμευτική. Τα κατώτατα αυτά ποσοστά Εδώ η πρόταση της Επιτροπής ήταν 56%, εγώ το έκανα 90%. Είμαστε ευρωβουλευτές και νομίζω ότι είναι δικός μας ρόλος να μιλήσουμε εξ των Χριστών, εξ αυτών που θα εμποφεληθούν από αυτή την κατάρτιση. Δεν θέλω να θυμώσει η Επιτροπή, αλλά πραγματικά εμείς είμαστε αυτοί που θα δείξουμε το δρόμο στο πρόγραμμα αυτό. Μετά από τρία χρόνια θα ξαναμιλήσουμε. Θα δούμε αν είχαμε δίκιο ή όχι. Εμείς θέλουμε μετά από τρία χρόνια να υπάρχει ευελιξία. Αλλά ευθύ εξ αρχής πρέπει να γίνει συγκεκριμένο το τι ζητάμε. Λεωνάρδο Νταβίντσι. Επαγγελματική κατάρτιση. Εγώ εδώ προτείνω ελάχιστη χρηματοδότηση 120%. 120% ο συνολικός προϋπολογισμός κανονικά θα αυξηθεί. Αυτό προτείνει η Επιτροπή. Συγγνώμη, 21% λέει η Πρόεδρος, το οποίο αρχικά είχε προταθεί να φτάσει στο 25% για το πρόγραμμα Λεωνάρτο Νταβίντσι όπως ξέρετε, θα χρηματοδοτηθεί στο μέλλον από το Κοινωνικό Ταμείο. Αν μπορείτε να μην τηλεφωνάτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα ήταν πιο ευχάριστο για μένα. Κύριε Κορέλ, μπορείτε να με ακούσετε. Το θέμα εδώ είναι οι διάφοροι τομείς κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των προγραμμάτων, αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές, να μπορούμε να αλλάξουμε. Παραδείγματο χάρη, το 2017, όταν γίνει η έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα γνωμοδοτήσει, θα κάνει κάποιες προτάσεις και βάσει αυτών των προτάσεων θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι δική μου πρόθεση και παρακαλώ πολύ να με ακούει η Επιτροπή. Δεν είναι δική μου πρόταση για όλους αυτούς τους τομείς να αποφασίσουμε εδώ στην κινητικότητα, στη συνεργασία, στις μεταρρυθμίσεις, να αποφασίσουμε εμείς πόσα χρήματα θα δοθούν για τη συνεργασία, για την κινητικότητα ή για τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του προγράμματος Κομένιος. Δεν θα σας το πω εγώ αυτό κύριε Κορέλ. Εγώ μπορεί να σας πω ποιο θα ήθελα να είναι το ποσό και από εκεί και πέρα το 2017 όταν γίνει μία αξιολόγηση μπορούμε να το αλλάξουμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βρεθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση για τον τελικό χρήστη. Όπως ξέρετε υπάρχουν εθνικές υπηρεσίες, οργανισμοί και φορείς. Η Επιτροπή ζητάει να υπάρχει μία μοναδική ανακράτος. Από την άλλη μεριά εδώ υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί και να έχει τη δυνατότητα να οργανωθεί όπως ε, είναι πιο χρήσιμο και πιο λειτουργικό για τις συνήθειες του κάθε κράτους. Η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει μόνο μία επιτροπή για κάθε πρόγραμμα. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ καλύπτονται πάρα πολύ διαφορετικοί τομείς για τον αθλητισμό, για τους νέους και για την κατάρτιση και για την ανώτατη εκπαίδευση. Προτείνω λοιπόν εγώ εδώ να παραμείνουμε σε αυτή τη δομή που προτείνει η Επιτροπή, αλλά να μπορέσει να υπάρξει ε, μια κατανομή ανά θέμα, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις και να παίξουμε τον ε, ε, ρόλο μας που είναι ένας ρόλος παρατηρητή σε ορισμένα σημεία, παραδείγματος χάρη για την επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικοί εταίροι. Και υπάρχουν οργανισμοί και φορείς, παραδείγματος χάρη, που μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο παρατηρητή στον τομέα, παραδείγματος χάρη, της εκπαίδευσης. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Λοιπόν, το Εράσμους για όλους δεν υπάρχει, είναι λανθασμένος τίτλος το Εράσμος είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι για όλους. Και θα πρέπει πραγματικά εδώ να ξαναδούμε κάποιες ονομασίες και τίτλους. Προτείνω λοιπόν εγώ στην έκθεσή μου για την διαβίου ε, κατάρτιση να παραμείνει ο τίτλος αυτό, αυτός είναι εξάλλου και η πρόταση της Επιτροπής. Ζήτησα Επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις. Η πρόταση ήταν yes, youth, education and sport. Yes. Τα τρία αυτά αρχικά. Το yes όμως το είχε χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος ε, σύλλογος, κάποια άλλα ένωση. Προτείνω λοιπόν να δεχτούμε το Yes Europe. Yes Europe. Πιστεύω ότι το 90% των μελών αυτής της Επιτροπής μπορούν να το δεχτούν. Σας ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι για την προσοχή σας και από εδώ και πέρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. First, ε, Τάκουλα. Κύριο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το ναι στην Ευρώπη, yes to Europe. Okay, I can continue. Θα συνεχίσω. Πολύ καλή δουλειά έκανε η Πρόεδρος. Θα κάνω λίγες παρατηρήσεις. Καταρχάς να πω ότι δουλέψατε πάρα πολύ έντονα. Και μετά τις συζητήσεις που κάναμε πάνω στο πρώτο σχέδιο με εθνικές οργανώσεις για το πρόγραμμα, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες. Ανησυχίες ότι αυτή η πρόταση μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες περιγράφοντας τις δράσεις. Και υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα καταστήσει την εφαρμογή δύσκολη. Ότι θα υπάρξουν δεκάδες ε, ξεχωριστές δράσεις και ότι αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό και ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το κόστος. Αυτές οι ανησυχίες, αυτή η φόβη εκφράστηκαν και από φιλανδού ενδιαφερόμενους. Από αυτούς κυρίως που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Μήπω το παρακάναμε τις λεπτομέρειες. Αυτό ήταν το θέμα που θέσανε. Αυτό ήταν η ανησυχία που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, Υπάρχουν γενικοί στόχοι και ειδικοί στόχοι. Υπάρχουν τομεακοί στόχοι επίσης. Και εκεί υπήρξαν ερωτήματα. Μήπως αυτό καταστήσει το πρόγραμμα περίπλοκο. Μήπως θα είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Μήπως θα είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε δείκτες για το πρόγραμμα. Αυτά είναι τα θέματα που ακούστηκαν και θα πρέπει να τα εξετάσουμε πριν να αποφασίσουμε τελικά για το πρόγραμμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σημαντικό να ακούμε τον κόσμο που θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Η αιτήσια έγκριση, άρθρο 27. Νομίζω ότι είναι μια πολύ επαχθής διαδικασία. Και επίσης τα άρθρα 21 και 22. Οι εθνικές αρχές στη Φιλανδία δεν θέλουν να επηρεάσουν τον τρόπο χορήγησης των θεωρήσεων. Και σε ό,τι αφορά την κατανομή της χρηματοδότησης. Επίσης, είναι πολύ σημαντική να δοθεί έμφαση ε, στην ε, γενική εκπαίδευση. Το 90% του προϋπολογισμού προβλέπεται στον κανονισμό. Αυτό θεωρήθηκε καλό. Τώρα, για τον τομέα του αθλητισμού. Πρέπει να αναφέρουμε ένα ελάχιστο ποσό για τα εθνικά γραφεία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, αν υπάρξουν περικοπές σημαντικά στο Συμβούλιο του προϋπολογισμού, ο προπολογισμό τελικά του αθλητισμού θα είναι τόσο μικρός που δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν υπάρχουν λιγότερα ε, χρήματα για τα εθνικά γραφεία σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα, με τη σημερινή περίοδο δηλαδή, θα είναι προβληματικό αυτό για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό. μιλάμε για το κομμάτι του αθλητισμού στο Εράσμους. Αν θέλουμε να έχουμε καλούς αθλητές, στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσουμε και λεφτά. Επίσης, το σύστημα εγγύησεων των δανείων. Δύσκολο το βλέπω. Τουλάχιστον εμεί στην Φιλανδία έτσι θεωρούμε. Και δεν είμαστε υπέρ αυτού του συστήματος. Θεωρούμε ότι είναι περίπλοκο. Πρόεδρε, αυτά είναι όσα μα λένε οι ενδιαφερόμενοι. Αυτοί που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Τα λένε καλόπιστα και επικοδομητικά. Γενικά, τους αρέσει το έρασμού. Αυτές είναι κάποιες μικροανησυχίε που ήθελα να σα διαμηνήσω. Εάν βρούμε λύση για αυτέ θα ήταν τέλειο.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 είναι πολύ καλύτερο αυτό το κείμενο από το προηγούμενο. Αυτό το σχέδιο κειμένου βελτιώνει το κείμενο της Κομισιόν. Και εγώ και η ομάδα μου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να λύσουμε το ειδικό κεφάλαιο, το θέμα του ειδικού κεφαλαίου για την νεολαία. Θα πρέπει να υπάρχει και ειδικό προπολογισμό. Να ξέρουμε ότι αυτός ο προπολογισμό θα πηγαίνει στην νεολαία. Πρέπει να το επιλύσουμε αυτό το θέμα, λοιπόν, του ειδικού κεφαλαίου για την νεολαία. Μην ξεχνάτε την πρόταση που συζητήσαμε στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Για αυτό το τρίτο τμήμα θα πρέπει να προτείνουμε ένα όνομα. Έχει προταθεί να χρησιμοποιήσουμε το όνομα «Η νεολαία αποφασίζει». Γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι είναι σημαντικό η νεολαία να αποφασίζει για το μέλλον της. Επίσης, το σύστημα ε, εγγύησεων των δανείων για σπουδές. Δεν έχουμε καταλάβει τι σκεφτόταν η Κομισιόν όταν το πρότεινε. Χρειαζόμαστε και καλύτερους ορισμού και καλύτερους κανόνες σε ό,τι αφορά αυτά τα δάνεια. Και χαίρομαι που θα οργανωθεί αυτή η συνάντηση με την Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μας τους σοσιαλιστές είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κριτήρια σε ό,τι αφορά αυτά τα δάνεια. Επίση όσοι δεν έχουν του πόρου. είναι σημαντικό να ξέρουν πού θα βρουν τα λεφτά για να σπουδάσουν. Όπως είπατε κι εσεί, κυρία Πρόεδρε. Δάνεια τα οποία δίδονται σε άτομα υπό το σύστημα κινητικότητας συχνά δεν επαρκούν. Το βασικό είναι να δίνουμε επαρκή δάνεια σε αυτούς που τα χρειάζονται για να σπουδάσουν. Επίσης θα πρέπει να προσαρμόζουμε τα δάνεια αυτά στο κόστος ζωής της χώρας όπου οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σπουδάσουν. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και την κατανομή του, το έχουμε συζητήσει διαμακρών στην Επιτροπή. Το 90% του προπολογισμού είναι ήδη κατανεμημένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό Αλλά εδώ μπορούμε να προτείνουμε ότι ίσως μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια η Κομισιόν μπορεί να υποβάλει μία έκθεση, ούτω ώστε και εμείς να μπορούμε ως Κοινοβούλιο να αλλάζουμε την κατανομή του προϋπολογισμού. Να είναι δυνατόν δηλαδή να γίνουν κάποιες αλλαγές όταν αυτό χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει το ότι έχει κατανεμηθεί το 90% του προϋπολογισμού. Η αίμα δεν είναι εδώ μαζί μας αλλά στη συνάντηση των σκιωδών συζητήσαμε και το θέμα του προγράμματος Ζαμονέ και το θέμα του αθλητισμού. Ε, συζητήσαμε την αναλογία αυτών των δύο προγραμμάτων στον προπολογισμό. Και μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι το τρίτος πυλώνας αυτού του προγράμματος. Ίσως θα μπορούσε να λάβει λοιπόν περισσότερα κονδύλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να το προβλέψουμε αυτό και να υποστηρίξουμε περισσότερο τον αθλητισμό, περισσότερα κονδύλια, Ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Αυτά από πλευρά μου και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Πιστεύω ότι θα βελτιώσετε ακόμα περισσότερο το κείμενο. Ο Μάρκος Κορέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την έκθεσή σα. Ελπίζω η Κομισιόν να μην προσβληθεί αλλά νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ πιο πλήρης, πολύ καλύτερη και πολύ καλύτερα οργανωμένη σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Τέλος πάντων, αυτό το ρόλο παίζουν εκεί οι δικές μας οι εκθέσεις. Θέλουν να βελτιώσουν την αρχική πρόταση. Νομίζω ότι το πετυχαίνετε και ικανοποιούμαστε όλοι. Νομίζω ότι πηγαίνει προς την κατεύθυνση που είχαμε υποδείξει και στις συνεδριάσεις της ε, Επιτροπής μας στο παρελθόν. Εξορθολογίζει το πλαίσιο καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε στην ε, διάθεσή μας ένα κεφάλαιο για την νεολαία, ένα για την εκπαίδευση κατάρτιση και ένα για τον αθλητισμό. Έτσι όπως παρουσιάζονται, στο κείμενο μου φαίνεται ότι γίνονται πολύ πιο εύληπτοι από τους αναγνώστες στο μέλλον. Άρα είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι γι' αυτό. Για τις agencies. Σας είχαμε πει να αφήσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν περισσότερες ε, υπηρεσίες και που λειτουργούν καλά, χωρίς υπερβολικά έξοδα και που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αποτελέσματα, ειδήσει, πληροφορίε σε όλη την επικράτεια, α πούμε, την εθνική, είναι σημαντικό να τι αφήσουμε να λειτουργούν και αυτό ήταν σημαντικό το ότι το πετύχαμε με το κείμενο. Είχαμε εκφράσει κάποιες ανησυχίες για το όνομα. Αυτό το Yes Europe, εντάξει, εμένα με πείθει. Νομίζω ότι είναι ένα όνομα αρκετά ελκυστικό. Νομίζω ότι είναι πιασάρικο για τις νέες γενιές. Νομίζω ότι περνάει ωραία και στα κοινωνικά δίκτυα. Νομίζω λοιπόν ότι και από αυτή την άποψη κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Υπάρχει όμως ε, ένα προβληματικό σημείο. Δεν είναι δικό μας λάθος. Ε, αυτό αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ εμπλέκονται πάρα πολλές ε, άλλες επιτροπές και παράλληλα προωθούνται ε, πολλές μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες και συζητούν οι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ας πούμε της γεωργίας κτλ. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τα τελικά ποσά, τα τελικά ποσοστά στον προϋπολογισμό. Πάντως, κατά τα άλλα, έχετε κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ, κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως και άλλοι σκιώδεις εισηγητές, και εγώ συμφωνώ και συμμερίζομαι τη λογική που διέπει την πρότασή σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και έτσι μεγάλη ορατότητα του προγράμματος προς τα έξω, αλλά και ευελιξία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση. Η πρόταση πάντως της Κομισιόν ξέρω ότι δεν αρέσει στους ε, εταίρους μας και ότι φοβούνται ότι το πρόγραμμα αυτό δεν θα γίνει γνωστό στους ε, Ευρωπαίους, γνωστός στους Ευρωπαίους. Για τόσο σημαντικά προγράμματα όπως αυτό χρειαζόμαστε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να μάθουν τα προγράμματα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και πρέπει να κάνει αυτή την προσπάθεια, εν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, από πλευρά μου, έχω δύο ανησυχίε. Θεωρώ ότι δεν βάζουμε αρκετή έμφαση στην ε, άτυπη και επίσημη εκπαίδευση. Και τι ρόλο δίνουμε στους φορείς της ε, επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης στο πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά τελώ εν συγχύση για να το πω έτσι. Τι θα παραμείνει στο πρόγραμμα για την ε, εκπαίδευση των ενηλίκων. Τη λογική του προγράμματος την καταλαβαίνω. Είναι εκπαίδευση και κατάρτιση διαβίου. Τι σημαίνει όμως ακριβώς αυτό. Δεν έχει ξεκαθαριστεί για μένα αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε στο θέμα των θεωρήσεων, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα. αν ε, διδαχθούμε αυτά που πρέπει να διδαχθούμε από το Erasmus Mundus, αν θέλουμε να γίνουν προσπάθειες προς τα εμπρός, πρέπει να λύσουμε το θέμα των θεωρήσεων. Να σας πω κάτι εμπαρόδο. Ήμασταν μαζί στη Δανία, στο Άρχους. Και θυμάστε αυτό το νεαρό Καμερουνέζο, ο οποίος επωφελήθηκε από αυτό το πρόγραμμα. Πραγματικά σας δείχνει τι πρέπει να καταφέρουμε με αυτές τις χώρες του Νότου. Αυτός ο άνθρωπος σας το δείχνει, έτσι πολύ παραστατικά ανάγλυφα, αν θέλετε. Τώρα, μια μικρή ανησυχία, που είναι μάλλον μεταφραστικό θέμα. Θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε. Ε, μιλάω για την τροπολογία 105 και το θέμα της κινητικότητας. Η κινητικότητα, εν προκειμένου, είναι η κινητικότητα των ε, φοιτητών και όχι των διπλωμάτων. Έτσι. Το βασικό είναι να επιτρέψουμε να κυκλοφορούν οι φοιτητέ. Παρότι βέβαια και η κυκλοφορία των διπλωμάτων τελικά δεν είναι ασήμαντο θέμα. Ε, αν συγκρίνω το γαλλικό κείμενο με τα άλλα, υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Πρέπει να διορθώσουμε το γαλλικό κείμενο. Ξέρετε τώρα ποια είναι η ανησυχία μου, η μόνιμη. Ξέρουμε όλοι μας ότι το Erasmus έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το λέω εγώ μόνο. Και αν λάβουμε υπόψη μας σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, καταλαβαίνετε πόσο επιτυχημένο ήταν το Erasmus. Είπατε σωστά, Πρόεδρε, ότι το Erasmus και προκύπτει και από τη μελέτη που έγινε, ότι το Erasmus δεν είναι για όλους, ε, είναι για αυτούς που μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν το έρασμος. Ε, αυτά τα δάνεια που, τα οποία αναφέρουμε, που αναφέρουμε συγγνώμη, είναι δάνεια σε κάποιους που μπορεί να τα συμπληρώσουν με δικά τους. Πρέπει να, πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα λοιπόν των τραπεζικών δανείων. Δεν πρέπει να δίνουμε ένα τέτοιο μήνυμα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ό,τι αφορά την εκπαιδευτική πολιτική, είμαστε εδώ για να δώσουμε προτεραιότητες, να στείλουμε μηνύματα, για να ευνοήσουμε τις καλές πρακτικές, να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Η προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουμε είναι να επιτρέψουμε στον κόσμο που προέρχεται από φτωχές οικογένειες, επίσης να έχει πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα. Και με αυτά τα δάνεια που προβλέπουμε, τα τραπεζικά δάνεια, δεν θα το καταφέρουμε. Το Yes μου άρεσε ήδη. Ε, το Yes for Europe μου αρέσει. Επίσης, μου αρέσει το μήνυμά του. Θα το συζητήσουμε μάλλον, φαντάζομαι, στην ομάδα μου αυτό το θέμα. Αλλά ο συμβολισμός που περνάει ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, ε, τον στηρίζουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, Πρόεδρε, για τη δουλειά που κάνατε. Είναι Yes Europe, όχι Yes for Europe το όνομα. Um, Herr Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η έκθεση πάντως ε, ήταν πάρα πολύ πλήρης. Ε, αποτέλεσε σωστή συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή μας θα πρέπει σοβαρά να κάτσει και να προβληματιστεί γιατί προχωρούμε με αυτό τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται τώρα για ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που ποτέ, που ποτέ έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να προσπαθήσουμε με αυτά τα οποία κάνουμε να σημειωθεί πιο ευρεία συνένεση. Βέβαια στην Επιτροπή μας υπάρχει μια μακρά παράδοση για τη συνένεση. Επίσης, νομίζω ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συνέντευξη στην Επιτροπή μας, σε τόσο πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση θα βρισκόμαστε έναντι του Συμβουλίου, όταν έρθει η ώρα. Επομένως, εδώ είναι η πρόταση της Κομισιόν, η δεδομένη, και οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι είναι θετική. Θα πρέπει επίσης, όπως έχουμε πει, να κάνουμε πιο ελαφρά, πιο ευέλικτα τα υπάρχοντα προγράμματα και το Συμβούλιο συμφωνεί προς τούτο. Άρα, από αυτή τη βάση να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει και να προσπαθήσουμε επομένω να αυξηθεί η προοικοδότηση προς τα προγράμματα. Αυτά πιστεύει η πολιτική μας ομάδα. Να δούμε για να θα αλλάξει θέση το Συμβούλιο πάντως. Για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι δάσκαλος, είμαι όμως δημοσιογράφος και έχω μάθει από τη δουλειά μου το εξή. Ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η αντίληψη. Δηλαδή, όσο καλές προθέσεις και να έχει κάποιος, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη το πώς θα αντιληφθούν οι χρήστε, α το πούμε, οι αποδέκτε τη του, αυτό το οποίο κάνει. Άρα θα πρέπει ακριβώς πάνω σε αυτό να προβληματιστούμε και να δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Χωρίς να ξεχνούμε, βεβαίω ότι τελικά θα πρέπει και η ανταπόκριση να είναι σωστή. Είναι σαφής στο κείμενο οι στόχοι σε σχέση με τους τελικούς ε, αποδέκτες και φυσικά αυτό δεν ήταν και εύκολο να γίνει. Μπράβο. Ε, έχουν μπει και στόχοι που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως είπε ο κύριος Στάκουλα. Και θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη ότι για κάποια κρατημέλη έχουμε υπερβάλλει κάπως, άρα θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο ισορροπία και να προχωρήσουμε προ την απλούστευση του προγράμματο, αλλά επίση να είμαστε και σίγουροι ότι οι χρήστε οι συμμετέχοντε στο πρόγραμμα θα έχουν αυτά που είχαν μέχρι τώρα. Άρα θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε σε κάποιο είδου συμβιβασμό. Ελπίζω θα τα συμφωνήσουμε εδώ στην Επιτροπή πριν πάμε για διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλάβει. Οπότε, για να δούμε τώρα. Ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής. Θα μελετήσαμε στην πολιτική μας ομάδα και όπως σας είπα συμφωνούμε και νομίζουμε ότι είναι αξιόλογη. Και να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή πλεύσης, ακριβώς για αυτούς τους τρεις τομείς, όπως τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τα λέει ο εισηγητής. Ταυτόχρονα επίσης, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τις, τις ίδιες ε, φίρμες, τις ίδιες μάρκες. Νομίζω πως μπορούμε να περάσουμε τις θέσεις μας στις διαπραγματεύσεις αν εδώ συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Και τελικά να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, Όσον αφορά τα, τα άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε αυτό, αυτά τα, τα δάνεια για τις μεταπτυχιακέ σπουδέ, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και φυσικά θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Συμφωνούμε, είναι θετικέ οι προθέσεις, αλλά πάντα ο διάβολο κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και άρα, να δούμε. με τέτοιο μέτρο αν θα μπορεί να αποδώσει. Το 56% που λέει ο συγκεκριτής ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Πάντως, θα πρέπει να παρακολουθούμε πόσα πηγαίνουν σε κάθε τομέα. 90% φυσικά είναι πάρα πολύ. Ε, ε, ναι, ε, όχι 90-75% θα έλεγα. τέλο πάντων θα πρέπει ίσω να βρεθεί η μέση οδό μεταξύ, ε, μεταξύ του ενό ποσοστού και του άλλου. Πολύ σωστά αναφέρεται αυτά τα έξι θεσμικά όργανα είναι όλα αξιόλογα άρα συμφωνώ με τα έξι και δεν νομίζω ότι κανείς ε, θα πρέπει να κολλήσει στα 6 αλλά γιατί και να υπάρξει μείωση και να πάμε στα δύο. Οπότε, όσον αφορά την πρόταση Yes Europe, είναι από τις καλύτερες προτάσεις που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Και θεωρώ ότι καθ' τον τρόπο θα μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα πάρα πολύ καλό οπότε και έτσι να προχωρήσουμε σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Euh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και εγώ και αυτή η πρόταση που μας κάνετε σήμερα με ευχάριστο τρόπο διαπιστώνουμε ότι έχετε εδώ καλύψει διάφορα. Πάρα πολλά από είπαμε στις συνεδρίες των σκιωδών. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων, ανάλογα με τη δράση, ανάλογα με, τον τομέα. Τα συζητήσαμε στην πολιτική μας ομάδα. Δεν καταλήξαμε σε συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά τέλος πάντων η κατανομή ανά πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέπετε ποσοστό. Αναρωτιέμαι τώρα, μήπως θα μπορούσαμε να δείξουμε ένα περιθώριο ευελιξίας 1-2% και έτσι να πάνε κάποια χρήματα για κάποιες δράσεις που δεν τις έχουμε ακόμα σκεφτεί. Κάποια στιγμή μπορεί κάτι να βγει. Και ίσως να μπορούμε λοιπόν να βάλουμε στην άκρη 1-2% για τις πράξεις που ακόμα δεν έχουν ανακύψει. Ας πούμε όσον αφορά Για την εγκατάλειψη του σχολείου δεν προβλέπεται ακόμα τίποτα. Οπότε μπορούν να προκύψουν διάφορα τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε για την ε, αναλφαβητισμό. Για τον αναλφαβητισμό επίσης δεν έχουμε πει τίποτα. Είναι παλιά προβλήματα αυτά. Οπότε ίσως θα πρέπει να υπάρχει αυτή το περιθώριο ευελιξίας. Τώρα σε αυτό το πρόγραμμα, ναι η πρόταση νομίζω ότι είναι αξιόλογη. Ίσως ο τίτλος είναι πολύ μεγάλος, έτσι όπως διατυπώνεται. Και ίσως να πρέπει να βρούμε κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Τώρα. Για ένα πρόγραμμα ειδικό που να στοχεύει στην νεολαία. Και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης εδώ καλύψατε το θέμα της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και το θέμα των θεωρήσεων. Ακριβώς για να μπορούμε να καλύψουμε και κάποιους από εκείνες τις χώρες. Επίσης έχουμε γι' αυτό το θέμα που με ενδιαφέρει τη συνεργασία με τις γειτονιάουσες χώρες της Μεσογείου. Άρα χρειάζεται εδώ ξεκάθαρη θέση και να είμαστε μπας συνεπείς με την πολιτική γειτνίασης που υπάρχει Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε ζωή μας σε αυτή τη συνεργασία. Να μείνει αυτή η μνήμα για τους ε, επιλέξιμους, για τους αποδέκτες του προγράμματος, φοιτητές, εργαζόμενοι, ενήλικες, όπως είπε η κυρία Βερζιά, στο πρόγραμμα που τρέχει ήδη, καλύπτονται αυτοί, αλλά όχι αρκετά γιατί εκτός από τους νέους υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο μεγάλοι που καταλήγουν άνεργοι και πρέπει να καταρτιστούν, να αποκτήσουν δεξιότητες για κάποια επαγγέλματα και κάποια καινούργια που βγαίνουν. Παρακάτω επίσης για το πρόγραμμα Ζώμονε άκουσα τη μόνη συνάδελφε και με ενοχλεί το ότι θα χρηματοδοτούμε θεσμικά όργανα. Προτιμώ να μείνει αυτός ο τίτλος αλλά να έχουμε ένα δίκτυο και να χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα μαθήματα, συγκεκριμένες σχολές που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Άρα όχι, όχι τις έδρες. Όσον αφορά τώρα αυτές τις εγγυήσει για τα δάνεια, πρόβλημα δημιουργεί το εξής. Υπάρχουν διάφορες χώρες που έχουν κάποια συστήματα περίπλοκα για τις υποτροφίες. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος επομένως να διαταραχτούν τα υπάρχοντα συστήματα. Κακό αυτό. Και επίσης είναι αλήθεια ότι Κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση στο αερασμό γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Άρα να βρεθεί τρόπος που να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα. Ίσως και αυτό να γίνει με, με δάνειο. Άρα να υπάρχει αυτή η εγγύηση για κάποια δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο κλπ. Οπότε να υπάρχει μια πλαισίωση συγκεκριμένη και με ένα τέτοιο σύστημα δανείων να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο έρασμος αν και δεν είχε τα χρήματα προς τούτο. Αυτά. Και σας ευχαριστώ και πάλι για το έργο σας. Και εγώ ευχαριστώ τον Πρόεδρος. Κύριο Πικάτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να μιλήσω για λογαριασμό της Emma Clarkin, η οποία ζητά συγγνώμη, αλλά έπρεπε να παραστής εργασίες του Φόρουμ Αθλητισμού στην Κύπρο και δεν μπορεί να είναι εδώ. δύσκολο να αλλάξει η δομή των προτάσεων της Επιτροπής. Οπότε και εμείς θεωρούμε θετικές αυτές τις προτάσεις. Όμως όσον αφορά την δομή του εγγράφου τελικά έχουμε κάποια δύσκολη να δεχτούμε, ε, να υπάρχει περισσότερη ευελιξία στα προγράμματα, να μειωθεί η γραφειοκρατία όμως αυτά που προτείνει η συγκεντρία και, και ε, τα ποσοστά αναδράση θεωρούμε ότι αυτό δεν θα αποτελέσει κίνητρο για την μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτά προσβεύει η κυρία Κλάρκιν και θέλει να το λάβετε υπόψη. Συμφωνούμε με την νομοδότηση, όμως θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για τον ευρωστεχνικό αθλητισμό. Αυτό δεν τονίστηκε αρκετά στην έκθεση και ιδίω τα κοινωτικά προγράμματα. Α πούμε έχουμε το Leader και επίση είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τι οργανώσει του θελοντικού αθλητισμού γιατί θα πρέπει να υπάρξει διεθνής αναγνώριση ως προϋπόθεση αυτό θα πρέπει να έρθει. αλλιώς ε, όλα τα χρήματα θα τα πάρουν ε, οι παλαιότερες πιο παραδοσιακές ε, οργανώσεις δηλαδή οι φορείς που τώρα πρόσφατα έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους δεν θα πάρουν τίποτα το πρόβλημα ε, αναφέρθηκε πριν Επομένω, κάποια χρήματα στον αθλητισμό. Έχουμε 380 εκατομμύρια, από τα οποία 338 πάνε στον αθλητισμό. Και εδώ έχει σταθεί η κυρία Κλάγκιν και λέει ότι αυτά τα δάνεια για τους ε, φοιτητέ θα καταστούν προβληματικά και άρα θα αποτελέσουν ε, πηγή ζημιών. Υπάρχουν ήδη συστήματα για την ενίσχυσή τους και επομένως το, το προτινόμενο σύστημα όταν κάποιος φοιτητής θέλει να πάει στο εξωτερικό θα δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα στην Ένωση. Επίσης ε, συμφωνούμε ε, κύριε Πακ ε, μαζί σας σε πάρα πολλά σημεία. Απλώς θα θέλαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά πιο, πιο στενά τις επόμενες μήνες. Κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι από απόψη της Επιτροπής είναι φιλόδοξο το σχέδιο, το πρόγραμμα. Απλοποίηση, επίσης ε, όσον αφορά την ε, ευελιξία που προτείνει, περισσότερη ευελιξία, κυρίως βέβαια για την Επιτροπή βλέπουμε να προτείνεται εδώ. Η πρόταση της Doris Pack είναι πολύ πιο σαφής κατά την άποψή μου όσον αφορά τη διατύπωση και όσον αφορά το περιεχόμενο. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια του σχεδιασμού και την ευελιξία που πρέπει να έχουμε, αυτή την αντίφαση, θεωρώ ότι έχει δίκιο η Doris Πακ όταν λέει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες δυνατότητες ευελιξίας με την έννοια ότι θα πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε ανάλογα με το τι συμβαίνει. Παραδείγματο χάρη, ξέρουμε σήμερα ότι λόγω της Αραβικής Άνοιξης κάποια από τα δεδομένα και τους αριθμούς που είχαμε σχεδιάσει και προγραμματίσει θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Θέλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς, όλοι οι οργανισμοί να μπορούν να προσαρμοστούν και την ίδια ώρα να υπάρχει και μια σχετική, αν θέλετε, ασφάλεια στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό. Να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ σχεδιασμού και ευελιξίας. Επίσης θεωρώ πολύ σωστό ότι εδώ κάνουμε μια παρουσίαση σαφή των διαφόρων ε, προγραμμάτων όσον αφορά παραδείγματο χάρη τη λεγόμενη άτυπη εκμάθηση, μάθηση, και αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει ιδιαίτερα να υποστηριχθεί. Ντόρις, μου αρέσει επίσης πολύ στην πρόταση το γεγονός ότι εμείς σαν Επιτροπή Πολιτισμού λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το ρόλο μας και ναι, μεν μιλάμε για ευελιξία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση κάποιων κονδυλίων, αλλά σαν Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίζουμε τον ρόλο μας που είναι ένας ρόλος ναι μεν συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θέλουμε να ακούγονται οι δικές μας απόψεις και το πολιτικό ειδικό βάρος που θέλουμε να θέσουμε σε ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Η στρατηγική του 2020 ο εξυγχρονισμός της οικονομίας μας που ελπίζουμε να γίνει με βιώσιμο τρόπο μας οδηγεί σε μια νέα θέση προτεραιοτήτων. Και καταρχήν η έννοια των φοιτητικών δανείων είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Αλλά αυτό το εργαλείο, αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει βεβαίως να γίνει με έναν τρόπο λογικό Δηλαδή, εάν σκοπός μας είναι στην Ευρώπη να υπάρχουν περισσότερα διπλώματα μάστερ, αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο εξισορροπημένο και με έναν τρόπο που να είναι θετικός για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το θέμα των θεωρήσεων επίσης θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να ρυθμιστεί και είμαι υπέρ του γεγονότος να διατηρηθούν τα κέντρα ζωμονέ οι δομές Ζωμονέ, γιατί έχουν αποδείξει ότι η εργασία που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι θετική και ότι μέχρι τώρα έχουν επενδυθεί σωστά ποσά για τον επιστημονικό τομέα και για την εκμάθηση συγκεκριμένων τομέων προς όφελος των νέων. Εμείς σαν πολιτικοί Ξέρουμε ότι η καλή πρόθεση βεβαίως είναι κάτι που μπορεί να εμπνεύσει. Όσον αφορά τον τίτλο λοιπόν Yes Europe, ναι, θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να δείξουμε θετικό πνεύμα, αισιοδοξία, Yes Europe, αυτά τα τρία αρχικά που συμπεριλαμβάνουν και τους νέους και την κατάρτιση και τον αθλητισμό. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος, μ' αρέσει αυτό το όνομα, αλλά βεβαίως αν υπάρχουν και άλλες ε, προτάσεις να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, η Πέτρα. Ευχαριστώ, Ντόρις. Θεωρώ πραγματικά ότι αυτή η κοινή ε, εργασία που οδήγησε στην ε, πρόταση, στην έκθεσή σου, είναι πάρα πολύ καλή. Η δική σου πρόταση σαφώς και αποσαφηνίζει το κείμενο της Επιτροπής γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται να έχει μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι δυνατότητες δίνει η Ευρώπη. Δίνεται ένας προσανατολισμός και μια περιγραφή πολύ πιο σαφής των διαφόρων προγραμμάτων και δυνατοτήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε σε πολύ καλή ε, οδό ακόμα και αν κάποια σημεία θα πρέπει να ξανασυζητηθούν και ελπίζω οι συζητήσεις με το Συμβούλιο να είναι ε, επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ε, μιλάμε για ένα μαύρο κουτί με λίγα λόγια και είναι πάρα πολύ δύσκολο γνωρίζοντας μόνο κάποια ποσοστά να θέσουμε κάποια όρια για όλες αυτές τις δράσεις. Και όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, παραδείγματος χάρη, στο Βερολίνο ακούσαμε πολλές επικρίσεις ότι δηλαδή θα μειωθεί το ποσό σε σχέση με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, ότι κινδυνεύουν να σταματήσουν κάποιες πολύ καλές πρωτοβουλίες. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Ε, τι είναι αυτά τα πραγματικά ποσοστά και πώς ανταποκρίνονται στους διάφορους τομείς. Συμφωνώ με αυτό που μόλις ε, ακούστηκε ότι εδώ μας δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα με τα δάνεια να βοηθήσουμε κάποιους νέους να κάνουν ένα μάστερ στο εξωτερικό. Ναι, πρόκειται για δάνειο. Ναι, πρέπει να αποπληρωθεί. Αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο δώσουμε ε, δυνατότητα σε κάποιους νέους που δεν έχουν αλλιώς τη δυνατότητα να το κάνουν. Εγώ όταν τελείωσα τις ποδές μου χρωστούσα 35.000 μάρκα. Ναι, δεν ήταν εύκολο να το αποπληρώσω. Από την άλλη μεριά δεν θα μπορούσα ποτέ με τις δυνατότητες που είχα τότε εγώ να κάνω αυτές τις σπουδέ. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε κάποιους νέους και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αποπληρωμή του δανείου, σε πόσα χρόνια, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να είναι υποφερτό για τους νέους αυτούς να τολμήσουν να πάρουν αυτά τα δάνεια, αλλά πραγματικά όλες αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να γίνουν με λογικό τρόπο, αλλά πραγματικά ας δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους νέους της Ευρώπης που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν αυτές τις σπουδέ. Ξέρετε ότι είναι μια επιπλέον ευκαιρία, μια επιπλέον δυνατότητα και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι η αποπληρωμή να είναι υποφερτή, να είναι λογική. Το Yes Europe, yes, εμένα μ' αρέσει. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά πρέπει να σας πω ότι ενθουσιάστηκα. Και ελπίζω τελικά να συμφωνήσουμε όλοι. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας παρουσιάσατε πολλές ιδέες στο κείμενό σας. Ειδικά για το Εράσμους για όλους. Συντάξτε μια θαυμάσια έκθεση που βελτιώνει πολύ την πρόταση της Κομισιόν. Το πρόγραμμα πηγαίνει πιο κοντά στους πολίτες. Μιλάει για δράσεις υπέρ του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας για τους πολίτες. Το θέλουμε. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προασπίσουμε και να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των πολιτών. Ε, η πρότασή σας είναι πιο κοντά στους πολίτες, λαμβάνει υπόψη περισσότερο τα συμφέροντά τους. Είναι λογικό εμείς να πολεμούμε για αυτά τα συμφέροντα και είναι λογικό να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε πρόταση βελτιώνει τις προτάσεις της Κομισιόν. Και η δική σας το κάνει. Τώρα, για την αυξημένη, ε, τον αυξημένο προϋπολογισμό για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Καλό είναι να έχουμε υψηλούς στόχους. Όταν ε, ήδη είναι γνωστό τι σημαίνει εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε πιθανές κρίσεις στο μέλλον αυτό, κρίσεις γενικά οικονομικές κτλ. Και, και η εκπαίδευση σίγουρα μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Σε πολλά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα. Ε, εδώ καλωσορίζω τα σχόλια των συναδέλφων που μίλησαν για προβλήματα εγκατάλειψης του σχολείου. Θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα στα κράτη-μέλη που καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο, αυτή την τάση. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πολυγλωσία επίσης, την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Και εδώ τα θερινά μαθήματα του Εράσμους μπορεί να βοηθήσουν. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους μειονεκτούντες, τις μειονεκτούσες ομάδες. Αυτό το ποσοστό το 90% είναι μια πολύ καλή αρχή για διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να μιλήσω επίσης για τον αθλητισμό για όλους. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά να δώσουμε προσοχή στον αθλητισμό για όλους. Φυσικά. Και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τους ε, νέους για τους μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν τα προγράμματα αθλητισμού να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι και για τους ερασιτέχνες. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε εθελοντικές δραστηριότητε για την νεολαία στον τομέα του αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά το Yes Europe, αυτή την ονομασία, το Yes, το ναι, αυτό είναι ένα καλό όνομα, μια καλή λέξη. Γιατί οι νέοι ε, τους νέους τους έλκουν, τους τραβούν οι απλές λέξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο κατάλληλο από το Erasmus for All, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι το Erasmus δεν είναι καθόλου για όλους. Επομένως, προτιμώ το Yes Europe. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ αυτών των πρωτοβουλειών σας, κυρία Πακ, και σας συγχαίρω. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πέκενοφ και κατόπιν η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είπατε πάρα πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Είναι εξαιρετική η έκθεση της κυρίας Πακ, θέτει στόχους κοινού ε, μεταξύ ημών και της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές όσον αφορά τους στόχους και πραγματικά θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ πιστική, αν θέλετε, παρουσίαση, μια σαφέστατη διάρθρωση, κατανομή της χρηματοδότησης, του προπολογισμού και μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική που θα οδηγήσει σε αυτούς τους στόχους. Μια στρατηγική η οποία τελικά οδηγείται από ένα σύγχρονο μάρκετινγκ θα έλεγα, Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και ενισχύεται εδώ ένας πολύ σημαντικός για μας τομέας όπως η επαγγελματική κατάρτιση. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι η διαβίου κατάρτιση είναι κάτι που ενισχύεται. Έχουμε ήδη επιτυχή αποτελέσματα και για άτομα που είναι πάνω από 40, πάνω από 50, το λεγόμενο LLL, Long Life Learning, διαβίου κατάρτιση, έχει δείξει, έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες και ότι είναι μια εξαιρετική βάση για να μπορέσουμε να απευθύνουμε αυτά τα μηνύματα και στους πολίτες και στους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορέτ έχει το λόγο από την Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Park. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πακ. Σα ευχαριστούμε επίση και για τόσο αξιόλογο κείμενο το οποίο ως συνήθως είναι πάρα πολύ πλήρες. Όπως θα γνωρίζετε δεν έχουμε καμία αμφιβολία και πάρα πολύ Είμαστε σίγουροι ότι προσέξατε τις δικές μας προτάσεις και εμείς επίσης προσέχουμε αυτά τα οποία λέτε. Πάντως, σαν καλός δάσκαλος είμαι επισμένος ότι θα πρέπει αυτά τα οποία διαβάζετε να διαβάζετε με κριτικό πνεύμα που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε την εκθέσή σας και θα πάρουμε, πάρουμε υπόψη στην πρότασή μας ε, και όσον αφορά τη συμφωνία με το Συμβούλιο είναι ότι για τα πιο βασικά είμαστε σύμφωνοι. Νομίζω συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα και μόνο πρόγραμμα και συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να δούμε την παιδεία, την νεότητα, τον αθλητισμό σαν τμήμα του ιδίου συνόλου να είναι επιμέρους δηλαδή το αυτή θα πρέπει να συνδέσουμε με την πολιτική ή τις πολιτικές μας το, το πρόγραμμα και επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απλή δομή και άρα συμφωνούμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής με αυτές τις τρεις δράσεις κλειδί θα εγκριθούν, θα περάσουν. Θα πρέπει επίσης να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της σαφήνειας. Γιατί αντιλαμβανόμεθα πως αυτά τα οποία λέει το Συμβούλιο και από την άλλη μεριά αυτά τα οποία εσείς λέτε, κυρία Πακ, τα οποία από ό,τι βλέπω τα εγκρίνουν τα μέλη της Επιτροπής, είναι το, ότι εμείς δεν έχουμε μια πρόταση με τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και σαφήνειας, οπότε θα πρέπει να το ξαναδούμε. Όπως σας είπα, έχω εμπειρία από την εργασία μου δασκάλου και άρα πιστεύω ότι τελικά θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες και θα τα βρούμε και δεν νομίζω ότι αν προσθέσουμε εδώ πέρα ε, ένα σωρό καινούριου στόχους θα κάνουμε τίποτα γιατί νέοι στόχοι θα είναι νέοι δείκτες και θα γίνει η ζωή πιο δύσκολη και για μας και για τους επιλέξιμους κάθε προγράμματος. Αντίθετα αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δούμε πιο λεπτομερώς το τι θέλουμε να κάνουμε με αυτές τις δράσεις κλειδιά, με την κινητικότητα και με τη συνεργασία. Όμως, δεν νομίζω ότι έτσι η ποσότητα θα φέρει περισσότερη σαφήνεια. Τέλος πάντων. Τελικά είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να αποσπάσουμε τα πιο ισορροπημένα αποτελέσματα. Επίσης και πάλι με αυτό το περίφημο κριτικό μου πνεύμα θέλω να δούμε τι θα γίνει με την κατανομή της προεκοδότησης, γιατί το είπαμε και το ξαναείπαμε ότι τελικά οι πολιτικοί θα αποφασίσουν για τα πιο βασικά που αφορούν το πρόγραμμα η Επιτροπή ουδέποτε το αμφισβήτησε και ούτε εγώ προσωπικά, όμως νομίζω ότι το να πάμε σε προετοιμασία πέραν του 90% κατά γνώμη μου αυτό θα αποτελέσει φραγμό σε δύο βασικά σημεία του προγράμματος. Πρώτα-πρώτα θα μειώσει τη δυνατότητα του να έχουμε διατομιακές δράσεις, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας και από την άλλη μεριά θα, έχουμε μικρό περιθώριο ελιγμών και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε σε ενδεχόμενες αλλαγές μεταξύ 14 και 20. Άρα να δούμε ποιο θα είναι το πιο σωστό επίπεδο ευελιξίας που θα αποφασίσουν από αυτού οι πολιτικοί. Και όπως είπατε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιον μηχανισμό αναθεώρησης και να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε ενδεχόμενε μεταβολέ και εν κατακλείδη να πω κάτι το οποίο δεν ελέγχθη μέχρι τώρα. Δηλαδή τι θα γίνει με το ετήσιο πρόγραμμα εργασία. Βλέπω στην πρότασή σα αναφέρεστε εδώ σε κάποια κατανομή αυτού του προγράμματο, κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Και εσεί θέλετε να έχει δύο τμήματα αυτό το πρόγραμμα και το ένα, όπως λέτε, θα πρέπει να αφορά τις και είναι τέλο πάντων να, να, να κρυθεί, να αποφασιστεί από τις κατανάθεση πράξεις εξουσιοδότηση πράξεις να δούμε όμως είναι αυτό συμβατό με το δημοσιονομικό κανονισμό Αυτά. Για γέννη και για τις λεπτομέρειες είμαι βέβαιος ότι στις αντίζεις που θα κάνουμε θα, τα πούμε μέχρι 6 Νοεμβρίου. Αλλά όπω σα είπα όλα αυτά σα τα είπα με κριτικό πνεύμα. Α, το τελευταίο. Όσον αφορά αυτή την εγγύηση δανείου για το μεταπτυχιακό υπάρχει γενικά σύγκληση απόψεων όχι ομοφωνία, σύγκληση απόψεων και ευρεία συνένεση για αυτή την ιδέα και αυτό δεν θα υποκαταστήσει τις ε, υποτροφίες θα τις συμπληρώσει θα τις επικουρεί ούτε θέλουμε να καταργήσουμε τα εθνικά συστήματα υποτροφιών άρα θα πρέπει να έχει το καινούριο σύστημα αρκετέ εγγύησεις που να σιγουρεύουν το ότι θα ωφεληθούν οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρόεδρε οι όρια προϋποθέσεις να δούμε το, το δεν θα καταλήξουν να μη δίνονται τα δάνεια αν είναι δηλαδή πάρα πολύ ευνοϊκή όρια για τους οφειλέτες. Τέλο πάντων το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, ένα από τα πιο σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν θα έχουν δύσκολο έργο γιατί ξεκινάμε ήδη από μια αφετηρία πάρα πολύ θετική καλά έφερνε στο πρόγραμμα, είναι δημοφιλέ, και τελικά να δούμε πώ θα έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα αυξάνει την ωφέλεια για του ε, ενδιαφερόμενους και αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι ούτε του Κοινοβουλίου μόνο, ούτε τη Κομισιόν, ούτε δικό. θα είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα ευχαριστώ. Βλέπω ότι έχουμε και τον ε, Κύπριο εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Äh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ε, Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Θα κοιτάξουμε όλες τις λεπτομέρειες με μεγάλη προσοχή και θα πάρουμε θέση. Πιστεύουμε ότι και προσβλέπουμε σε μια πολύ θετική συνεργασία και μαζί σας και με όλους τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και εγώ γιατί βασίζομαι πραγματικά στο Συμβούλιο. Έχω σημειώσει τις προτάσεις του Συμβουλίου. Τις έχω ενσωματώσει, όπως είδατε, στο κείμενό μου και ξέρω ότι ελπίζατε ότι εμείς θα προτείνουμε αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον να μας υποστηρίξετε όμως. Μιλάτε και τόσο καλά γερμανικά που πραγματικά είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσετε. Κύριε Κορέλ, δεν άκουσα τίποτα για τον τίτλο. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει αυτός ο τίτλος. Καλός δεν είναι. Ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Και τώρα περνάμε σε ένα σημείο. Θέλετε να πείτε κάτι. Ε, δεν σας ακούσαμε. Το γεγονός ε, ότι δεν είπα τίποτα δεν σημαίνει ότι μ' αρέσει κιόλα. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Και πολλοί ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι πρέπει να βρούμε ένα ωραίο τίτλο. Θέλουμε ένα καλό όνομα για το πρόγραμμα που πείθει τους πολίτες και να είναι εξίσου καλό με το όνομα που έχουμε και σήμερα. Αχ, κύριε Κορέλ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, αν ήσασταν ειλικρινείς, θα λέγατε ναι, περιπτώσει, περιμένετε να δείτε τι θα πει και η κυρία Βασιλείο. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολύ τεχνικό το θέμα, δεν αναφέρθηκα στα τεχνικά κομμάτια, όπως παραδείγματο χάρη την κατεξουσιοδότηση, της κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, εδώ θα πρέπει να υπάρξει κοινή ψηφοφορία με άλλους φορείς στο πρόγραμμα. Ναι, Θέλουμε λοιπόν εδώ να παραμείνουμε στην θέση της νομικής υπηρεσίας. Δεν θα μπορέσω εδώ να ακολουθήσω την πρόταση της Επιτροπής. Έχω υποβάλει τροπολογία και είμαι 100% σίγουρη ότι ακριβώς η ίδια συζήτηση θα ακολουθήσει για όλα τα προγράμματα. Πρόκειται για την διαφορά μεταξύ των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των άλλων και βεβαίως Ξέρω ότι κάποια στιγμή εδώ θα πρέπει να υπάρξει μία λίγο πιο τολμηρή στάση μεταξύ ημών, μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Κύριε Κορέλ, πιστεύω ότι δεν θέλετε να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Εγώ πραγματικά δεν άλλαξα τίποτα, τίποτα τα τρία σημαντικά θέματα όπως τα έχετε θέσει. Τις τρεις κατευθυντήριες γραμμές, τη συνεργασία, την κινητικότητα και τις ε, μεταρρυθμίσεις. Πραγματικά, πραγματικά. Το μόνο που έκανα ήταν ότι τα παρουσίασα με έναν πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Τίποτα άλλο. Αυτός που θα πάρει αυτό το πράγμα, το Yes Europe, να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Και αν κάποιος πραγματικά θέλει να μπει στις λεπτομέρειες, να καταλαβαίνει. Εγώ πραγματικά με αφορά να καταλάβει ο πολίτης, όχι η διοίκηση. Και δεν νομίζω ότι μειώνουμε την απλοποίηση, αν απλά και μόνο πριν διαβάσει κανείς το κείμενο, μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα αν το λέμε ήδη εκ των προτέρων με ένα ξεκάθαρο τρόπο, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν που δεν έχει ακόμα διαβάσει το κείμενο να το διαβάσει. Δεν είμαι κατά της απλοποίησης και δεν αφορά την απλοποίηση αυτό που σας λέω. Όποιος κάποιος, δεν, κάποιος αν κάποιος δεν θέλει την απλοποίηση, ας το πει. Εδώ δεν μειώνουμε την απλοποίηση, τις απλοποιημένες διαδικασίες. Κύριε Κορέλ, αν διαφωνείτε, μπορείτε να έρθετε να με δείτε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Επίσης, για τον αθλητισμό. Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει αθλητισμός. Στο YES υπάρχει το youth, η νέη, education, η κατάρτιση, η παιδεία και S, το sport, ο αθλητισμός. Απλώς έχουμε πάρα πολύ λίγα χρήματα για τον αθλητισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να βρούμε κάποια χρήματα από αλλού. Ναι, αλλά το, ο προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση. Τώρα, αυτό που είπατε όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, κύριε Τάκουλα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είπατε. Δεν κατάλαβα. Αλλά αν συζητήσουμε διμερώς, ίσως καταλάβω. Κυρία Βαντάλοβα, σας ευχαριστώ για τα περισσότερα από όσα είπατε. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα τα είχαμε συζητήσει και είχαν ληφθεί υπόψη. Το θέμα τώρα των ποσοστών για τον αθλητισμό, τι να σας πω, δεν είναι ο συνάδελφος από την Κυπριακή Προεδρία, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πραγματικά κάτι μπορούμε να κάνουμε, γιατί και για τους νέους και για την κατάρτιση πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη επεξεργασία η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο συγκεκριμένα ποσοστά. Καταλαβαίνετε ότι εγώ σαν εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδας και σαν εισηγήτρια συμφωνώ με τις προτάσεις που έκανα και κάτι που είπε ο κύριος Κορέα. Πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Εγώ συνεργάζομαι στενά με τον κύριο Μπέγκε και σίγουρα και με τον κύριο Μπέγκε, ο οποίος την τελευταία διαπραγμάτευση για, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου πέτυχε αύξηση ποσού για μας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πιστεύω ότι και εγώ αλλά και εκείνος θα πολεμήσουμε ακόμα. Ακόμα και ο κύριος Σούλτς μου είπε ότι μίλησε με την καγκελάριο, με την κυρία Μέρκελ, η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τον τομέα αυτό και σίγουρα κάτι θα γίνει στο μέσο πρόθεσμο. Τι να σας πω, αν αυτά που μου είπε τα κάνει κιόλα τόσο το καλύτερο. Κύριε Λόκεγκαρτ, κύριε Δάκουλα, σίγουρα πρέπει κάποια σημεία να τα ξανασυζητήσουμε. Το πρόβλημα τώρα είναι τι χρηματοδότηση θα πάρουμε για αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό δεν εξαρτάται από το πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Αν θα το παρουσιάσουμε όπως εμείς το παρουσιάσαμε ή κάπως αλλιώς. Εξαρτάται από το αν αυτό το πρόγραμμα είναι φιλικό προς το χρήστη, αν θα χρησιμοποιηθεί. Και μέχρι το 2017 και το λέω αυτό στην Επιτροπή, δεν θα έχει αλλάξει τόσο πολύ πια η Ευρώπη και ο κόσμος έτσι ώστε να έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Δεν σας ανέφερα όλα τα οποία γράφει το κείμενό μου, αλλά σαφώς και οι γειτονικές χώρες, οι όμορες χώρες οι χώρες όπου έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη συμπεριλαμβάνονται. Δεν το είπα, αλλά εννοείται. Και υπάρχουν επίσης και τρίτες χώρες. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τρίτων χωρών και γειτονικών χωρών, όμορων χωρών. Και το πρόγραμμα, επειδή ακριβώς περιέχει τόσες τόσο περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Αλλιώς τελικά θα περιορίσουμε ακόμα πιο πολύ τα ποσά που διαθέτουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν και είναι σαφέστατο, ήταν για μένα αυτονόητο, γι' αυτό και δεν το ανέφερα, ότι οι γειτονικέ χώρε είναι εντό, όπω είναι εντό και οι χώρε που βρίσκονται στην προενταξιακή διαδικασία και οι τρίτες χώρες. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν αναφέραμε τους νέους, αναφέραμε την κατάρτιση. Αν θεωρείτε ότι κάτι λείπει από την δική μου διατύπωση, μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογία. Τώρα, η διαβίου κατάρτιση. μετά τα 45. Μετά τα 45 είναι το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και λειτουργεί και το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί. Παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των seniors. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ πετυχημένο θα έλεγα σαν πρωτοβουλία και γι' αυτό και ήθελα να το αναφέρω. Όταν μιλάμε για κατάρτιση ενηλίκων, βεβαίως είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορεί όμως αυτό βεβαίως να αντικαταστήσει αυτό που προϋπάρχει, δηλαδή την ανώτατη εκπαίδευση ε, και την εκπαίδευση των νέων. Κύριε Μιγκάτσικη, δεν είστε εδώ, δεν χρειάζεται να απαντήσω. Κυρία Τρίπελ, με υποστηρίξετε σχεδόν σε όλα. Τώρα για το ζώμο ναι. Το ανέφεραν αρκετοί ομιλητές. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα προγράμματα αυτά, τα Ινστιτούτα αυτά, στη Φλωρεντία ή στο Άμστερνταμ, στη Μάστρικ, στο, στο Μάστρικ βρίσκονται δεν είναι Ολλανδικά Ινστιτούτα. Πρόκειται για φοιτητέ από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που σπουδάζουν εκεί. Πρόκειται για φοιτητέ εντός αλλά και εκτός Ευρώπης και πρόκειται για μια πολύ ισχυρή βάση. Δεν πρέπει αυτό να το αποδυναμώσουμε. Αυτά τα Ινστιτούτα εργάζονται όπου και να βρίσκονται στην Ευρώπη έχουν μια ακτινοβολία ευρωπαϊκή και παγκόσμια, διεθνή. Κυρία Μπενάβατου, μιλήσατε για τους καθηγητές. Οι καθηγητές ζώμων, στο, στα Ζώμονε θα παραμείνουν. Οι έδρες αυτές θα παραμείνουν. Προσθέτουμε επιπλέον αυτά τα Ινστιτούτα. Απλώς ε, η πρόταση για να συμπεριλάβουμε και άλλα Ινστιτούτα και άλλα Ιδρύματα, εδώ δεν αρκεί ο προπολογισμό φοβάμαι. Τώρα, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τα ποσοστά, λέτε, είναι πολύ χαμηλά. Αν αυτή η αύξηση που προτείνει η Επιτροπή γίνει πραγματική, ναι, θα ξεπεράσουμε το 25%. Αλλά αυτό είναι η προϋπόθεση, να υπάρχει η αύξηση. Ό,τι, αν θέλετε, έγινε μέχρι τώρα στο Λεωνάρντο, θα χρηματοδοτηθεί από εδώ και πέρα από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Μιλήσατε για τον αθλητισμό, κύριε Μάτουλα. Ναι, θα βελτιωθεί το πρόγραμμα, τουλάχιστον βάσει της δικής μου πρότασης βελτιώσαμε τη διατύπωση και εδώ ακολουθήσαμε αυτά που επιθυμεί το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτή είναι και η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτά άκουσα από όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υποστήριξή σας, για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας και ήθελα να σας πω ότι πολλά από αυτά που είπατε τα έχω ακούσει τους τελευταίους μήνες και τα έχω συμπεριλάβει. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας πω Κοιτάξτε λίγο και τις δικές μου προτάσεις και μην κάνετε την ίδια πρόταση στο κείμενο της Επιτροπής, αν το έχω εγώ συμπεριλάβει στη δική μου πρόταση. Κοιτάξτε περίπου τι έχω κάνει για να είμαστε σε συνδυασμένες παρατηρήσεις και προτάσεις. Τι να σας πω, είπα, ξαναείπα, επανέλαβα, όπως σας είπα ήμουν καθηγήτρια, ελπίζω η Επιτροπή να με κατάλαβε και να έχουμε μια θετική συνεργασία από εδώ και πέρα. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 11 θα μας παρουσιαστεί εδώ η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για πολιτιστικά έργα. Εμάς διαρκώς μας λένε γιατί δεν κάνετε αρκετά, γιατί είστε τόσο περιορισμένοι στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά έργα. Και μας τίθεται πολλέ φορέ και το ερώτημα τι δυνατότητε υπάρχουν για χρηματοδότηση μέσω των διαρθωτικών ταμείων. Όποιο θέλει να βγει από την αίθουσα παρακαλώ πολύ μπορεί να βγει τώρα. Γιατί αλλιώ κάνετε πολύ θόρυβο, δεν ακούμε. Just a moment. Who is the lady? You? Okay. Good morning, everybody. Καλημέρα. Okay. Please, eh, Madame Valentina Montalto, you have the floor. κυρία Βαλεντίνα Μοντάλτρο, έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη μελέτη και να σας δείξω πού βρίσκεται ο πολιτισμός ε, στην τρέχουσα πολιτική και στη μελλοντική πολιτική. Ε, μας ζητήσανε αυτή την ε, μελέτη από το ΚΕΑ. Ε, ο στόχος είναι να δώσουμε κάποιες συστάσεις και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα διαρθωτικά ταμεία για τον πολιτισμό υπό την τρέχουσα πολιτική και τη μελλοντική πολιτική μέχρι το 2020, 14-20. Ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της μελέτης με τον πολιτισμό. Αυτό σημαίνει πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες. Δηλαδή, καλλιτεχνικός κλάδος, ε, οπτικοακουστικός κλάδος κτλ. Ο πολιτισμός είναι και η παραγωγή πολιτιστικών έργων, δηλαδή μουσική, οπτικοακουστικά υλικά και δημιουργικός κλάδος ε, σημαίνει ο κλάδος, η κλάδη μάλλον, όπου ο πολιτισμός ε, είναι, ας πούμε, χρησιμοποιείται για να παράγουμε κάποια έργα, αρχιτεκτονική, σχέδιο κτλ. Ε, έχουμε κάνει, λάβει υπόψη μας την οικονομική επίπτωση του κλάδου. Ε, επηρεάζει πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, περίπου 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης δίνει. Ο κύκλος εργασιών είναι 654 εκατομμύρια και έχουμε και 1,4 εκατομμύριο εταιρείε. Ο πολιτισμός δεν συνεισφέρει μόνο στην οικονομία άμεσα, αλλά συνεισφέρει επίσης και στην ε, κοινωνική καινοτομία. Αλλάζουν τα μυαλά στην Ευρώπη και στον πολιτισμό και στην, στο δημιουργικό, στους δημιουργικούς κλάδους και στις σχετικές πολιτικές. Ε, υπάρχει η ατζέντα για τον πολιτισμό που θεωρείται ο πολιτισμός εργαλείο για τη δημιουργικότητα, για τον πολιτιστικό διάλογο αλλά και για τις διεθνείς σχέσεις. Επίσης, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση για την κοινοτομία. Λαμβάνουμε υπόψη μας και τις επενδύσεις στο σχέδιο και στις δημιουργικές βιομηχανίες. Και επίσης έχουμε ε, το πρόγραμμα Έξυπνη Ανάπτυξη από το 2010 και μετά. Ο πολιτισμός θεωρείται ως ελκυστικό στοιχείο για τις πόλεις και τις περιοχές μας και επίσης η καινοτομία και η δημιουργικότητα συνδέεται μέσω του πολιτισμού. Υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Καλλιτεχνικών Κλάδων. Ε, έχουμε μια έτσι επιχειρηματική ματιά και προσέγγιση για τον κλάδο. Ε, υπάρχει και η νέα Γενική Διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων που ασχολείται ε, με αυτά τα θέματα αλλάζουν τα μυαλά, αλλάζει το μοντέλο. Ε, θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η αλλαγή. Έχουν δοθεί 6, δισεκατομμύρια στον πολιτισμό. Ίσως δεν αρκούν, γιατί είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή το ποσά που ξοδεύουμε για τις, για τις καλλιτεχνικές βιομηχανίες, τους καλλιτεχνικούς κλάδους. 2007-2013 και επίση θα πρέπει αυτό να το δούμε σε σχέση με τι προτεραιότητε τη πολιτική συνοχή. Αν τώρα ρίξουμε μία ματιά ει ε, την πολιτική αυτή για, για τον πολιτισμό, ε, εμφανίζεται, ε, προκύπτει και στον κανονισμό του Ταμείου Ανάπτυξη και στι δράσει επενδύσεων. Όμω παρόλα αυτά η βασική παραπομπή στον πολιτισμό συνδέεται περισσότερο στον αφορά την κληρονομιά. Και αν ρίξετε μία ματιά επίση, σε αυτές τις κατευθυντήριες κοινές γραμμές θα διαπιστώσετε ότι και εν προκειμένου ε, καλύπτεται ο πολιτισμός, το πώς θα επενδυθεί εκεί, επομένως βλέπουμε ότι είναι soft location factor. Και επομένως έχουμε εδώ πέρα ε, και κάποια δημιουργία κινήτρων το οποίο είναι θετικό. Όμως αυτό το οποίο λείπει είναι μια παραπομπή, μια αμνία στο καινούριο περιεχόμενο του, του, πολιτισμού. Δηλαδή ότι είναι μέσω καινοτομία, ότι είναι ε, μια πηγή για να απτυχθεί η νέα οικονομία. Και όλα αυτά ε, αναλύεται. Έχουμε εδώ πέρα διάφορες ε, ε περιπτώσεις, διάφορες υπόθεσεις μελέτης και όλες αυτές μας δείχνουν ότι οι πόλεις, οι περιφέρειες και κάποια κράτη-μέλη είναι είναι, είναι, δεν καλύπτονται από, από, από έναν ευρύτερο ορισμό. Και άρα θα πρέπει, ε, να, κοιτάξτε, το Βερολίνο είναι ένα πάρα πολύ 38 παράδειγμα. Είναι μια δημιουργική πόλη σε εισαγωγικά. Και πάνω από ένα δις έχουν επενδύσει μέσω των διευθυντικών ταμείων, τόσο ώστε να, να κάνουν αυτή τη, τη, τη δουλειά και έχουν μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης όπως το λένε το Τσούκουμ του Μπερλίν και επίσης ε, στη Φιλανδία, άλλο παράδειγμα, έχουμε και εκεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εδώ πέρα το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε συγχρηματοδότηση προκειμένου με το κοινωνικό ταμείο. Και ε, αυτό είναι κάπως ε, σπάνιο να έχουμε για αυτό τον τομέα τέτοια προγράμματα που να συμμετέχει το κοινωνικό ταμείο και το Υπουργείο Παιδείας τελικά ε, συνεργάστηκε και έπεισε το Υπουργείο Οικονομίας να υπάρξει ένα ad hoc πρόγραμμα για τον τομέα και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, νέου τύπου επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει για την δημιουργική Εστονία, όπως λέμε. Θα το δείτε και στην επόμενη διαφάνεια. Επίσης έχουμε και ένα νέο προϊόν, ένα νέο πρόγραμμα που λέγεται Creative Spin ή Urbact. Ναντ. Γιατί ασχοληθήκαμε με την πόλη αυτή, γιατί τα πήγαν πάρα πολύ καλά αξιοποιώντα τα κονδύλια των διαστατικών ταμείων. Ε, έχει βέβαια παρελθόν ένδοξο βιομηχανικό η πόλη, αλλά στο τέλο τη δεκαετία του 80 ε, υπήρχε πρόβλημα με τα ναυπηγεία και η πρόκληση ήταν το πώς θα αναζωογονηθεί ο βιομηχανικό τομέα και πώ θα μπορέσουν ε, να ελκύσουν σε αυτή την περιοχή και τουρίστες αλλά και τον τόπιο κόσμο. Είναι ένα νησί κοντά στο κέντρο της πόλης ε, και ξεκίνησε πριν από μια εικοσαετία ε, περίπου ε, η, το, μια, μια ενασχόληση της περιοχής αυτής των καλλιτεχνών, θέατρο κλπ. Υπήρξε το, ένα φεστιβάλ και όπως είπαμε διάφοροι καλλιτέχνες προσπάθησαν να αναδομήσουν, να, να, δώσουν καινούργια εμφάνιση ε, εκεί στην, στην περιοχή αυτού του λιμανιού. Οπότε είχαμε επανέβαση ε, ε, καλλιτεχνική, ε, δημιουργικές, δημιουργικές εταιρείες προσέξανε και το οικοσύστημα. Έχουμε τώρα βέβαια και την αρχιτεχνική σχολή που βρίσκεται εκεί και η σχολή καλοτεχνών εκεί πρόκειται να εγκατασταθεί. Ε, τώρα, η πολιτική υποστήριξη για τον πολιτισμό σαν μέσο αναζωγόνης της περιοχής ήταν και αυτό κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και ο σημερινός πρωθυπουργός, ξέρετε, είναι ο πρώην δήμαρχος της πόλης. Οπότε και υπήρξε υποστήριξη πολιτική προς την, την πόλη για να δοθεί καινούργια όθηση στην οικονομία και στην συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Οπότε τώρα δεν είναι απλώς μια πόλη που περνάει κανείς σαν ενδιάμεσο σταθμό, σαν transit που λέμε. Είναι, είναι τουριστικός προορισμός. Και επίσης τώρα παίξει καινούργια εικόνα, καινούργιο προφίλ πολύ. Βλέπετε εκεί δεξιά. Δεξιά έχουμε αυτόν τον ελέφαντα. Αυτό το, το ονομάζουν μηχάνημα για τις τέχνες. Which is a medium-sized but have been found also in smaller cities. Και σε μικρότερες πόλεις όπως το Ταρτού έχει γίνει το ίδιο. Πόσο μεγάλο ενδιαφέρον πιο μικρή πόλη. Αυτές οι πολιτιστικές δημιουργικές βιομηχανίες αυτό ήταν μέρος του προγράμματος Δημιουργική Εστονία. Τα διευθυντικά ταμεία συγχρηματοδότησαν και ο στόχος, η πρόκληση εκεί στο Ταρτού ήταν το πώς θα ελκύσουν ή πώς θα κρατήσουν. 100.000 είναι οι κάτοικοι και 20.000 από αυτούς είναι θεατές. Άρα έγινε και προσπάθεια να στηριχθούν οι νέοι επιχειρηματίες. Να τους δώσουν ένα λόγο για να μην εγκαταλείψουν την πόλη. Τέλος, το Creative Spin. Νέο πρόγραμμα. Και ο στόχος του προγράμματος είναι το πώς θα συνδεθούν με τις ε, δημιουργικές τέχνες του Βερολίνου και τους άλλους τομείς της οικονομίας. Άρα είναι κάτι που έχει σχέση με αυτές τις ε, δημιουργικές πολιτικές. Ε, εδώ βλέπετε τη σχέση δηλαδή μεταξύ καινοτομίας και πολιτισμού. Βλέπουμε εδώ πώς γίνεται η διαχείριση, η διακυβέρνηση και ο στόχος, ο σκοπός είναι να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος ούτως ώστε ο πολιτισμός και άλλοι κλάδοι της οικονομίας να διασυνδεθούν και επίσης ε, ο πολιτισμός να αναζητήσει νέες αγορές, νέους αποδέκτες και τελικά έχουμε πάντα υπόψη μας τις μελλοντικές πολιτικές αλλά κυρίως τη μελλοντική οικονομία. Ρίξτε τώρα μια ματιά για το τι γίνεται στη νέα πολιτική της συνοχής. Και πιο συγκεκριμένα να δούμε την πρόταση της Επιτροπής. Έχει νέα, διαφορετική αρχιτεκτονική, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Απλώς σας επισύρω την προσοχή στο τι ισχύει σε σχέση με αυτές τις προτάσεις. Έχουμε τον κανονισμό του Ταμείου Ανάπτυξης και λέμε ότι θα πρέπει η πολιτική κοινωνία να προστατεύεται και να προωθείται κλπ. Το κοινό στατικικό πλαίσιο, καλύπτει τον πολιτισμό, για τις ΜΜΕ, για τις δημιουργικές βιομηχανίες, όλα αυτά έχουν σχέση με τον πολιτισμό αλλά και τις διαπολιτιστικές δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, τα πολιτιστικά δεν είναι θεματική προτεραιότητα για τη νέα πολιτική συνοχή. Στον δε του ERDF η παραπομπή στα πολιτιστικά παραμένει. Αλλά δεν αναφέρονται οι υποδομές, οι δημιουργικές βιομηχανίες σχετικά με τα πολιτιστικά. Δεν πρόκειται περί κανονισμού. Είναι ένα σχέδιο κανονισμού και υπόκειται στη διαδικασία αναθεώρησης τώρα από την Επιτροπή. Πάντως αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για κρατημέλη και περιφέρειες είναι ότι τώρα δίνεται με αυτή τη νέα πολιτική η ευκαιρία να διασυνδεθούν αυτές οι επιχειρήσεις με τις ευφυείς στρατηγικές εξειδίκευσης, smart specialization strategies. Οπότε και σε επίπεδο θα συνδεθεί αυτό το όραμα με τον πολιτισμό. Και αυτοί σε καινούργιε στρατηγικέ είναι προπόθεση ούτω ώστε κανεί να μπορεί να προσφύγει στα διαρθρωτικά ταμεία. Άρα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Οπότε, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι βέβαια και υπάρχει μια στροφή στην πολιτική προς ε, μια συνολικότερη κατανόηση των πολιτιστικών. Και έχουμε τις διάφορες υποθέσεις μελέτες όπου ο πολιτισμός δεν θεωρείται σαν ένας ακόμα τομέας αλλά σαν, σαν ε, πηγή. Σαν πηγή για ανάπτυξη στρατηγικών και ε, κυρίως πολιτικών που βοηθούν την καινοτομία. Το Creative Estonia, τη Δημιουργική Εστονία, επίσης το πρόγραμμα για την Νάντι που δεν θα υπήρχαν αυτά ούτε και καν και το του Βερολίνου αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη των διεθνών ταμείων και κάθε φορά ε, βλέπουμε πώς, τι, τι αντίκτυπος υπάρχει στην τοπική στήριξη στον να σου, δηλαδή κάθε, κάθε χώρο σε αυτό το πρόγραμμα και το Ιντερέ και το Ούρμπακ το πρόγραμμα επίσης ε, είναι, και αυτά πάρα πολύ σημαντικά το Interreg τα καλύπτει όλα τα, προηγούμενα προγράμματα για τις πόλεις που είπαμε, αφορούν ε, ε, όχι γραφειοκρατία, αλλά ανταλλαγή εμπειριών, ε, εμπνεύσεων, όμως όλα αυτά αντικατοπτρίζονταν μέρη μόνο στο έγγραφο για την πολιτική ε, 2014-2020 οπότε και έχουμε διατυπώσει κάποιες ε, συστάσεις. Πρώτα-πρώτα, ορισμός των πολιτιστικών, ορισμός του πολιτισμού να θεωρηθεί ως πηγή βιώσιμης ανάπτυξης. ανάπτυξης. Και να σας διαβάσω τώρα ένα κομμάτι από μια μελέτη που έγινε πέρσι. Αναφέρεται ακριβώς τον πολιτισμό σαν αηφόρο ε, ανάπτυξη και ότι η πολυμορφία των πολιτιστικών δεν αφορά την, την μορφή και τον τύπο, απλώς το πώς θα περιφορήσουμε το, τον, την ατομική ικανότητα της ανανέωσης. Ο πολιτισμός είναι πηγή βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλει ε, στην ανάπτυξη της Ευρώπης και επίσης ε, οφείλει και τις μέλους της γενναίας. Επομένως, είναι η ιδέα του πώς θα διασώσουμε, πώς θα συντηρήσουμε για το παρελθόν, αλλά και κυρίως για το μέλλον της Ευρώπης τον πολιτισμό. Άρα έχουμε εδώ πέρα μια νέα θεματική προτεραιότητα που να καλύπτει τον πολιτισμό μετά από τον νέο ορισμό. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει αυτή η προτεραιότητα η καινούργια να περιληφθεί στις προτεραιότητες που έχουν σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη για τους λόγους που προανέφερα. Κατόπιν έχουμε επίσης κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς τα πολιτιστικά θα, θα περάσουν σε όλες τις πολιτικές σε σχέση με την ανάπτυξη, την μη τεχνολογική, την κοινωνική ανανέωση, την ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων σε, και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και πώς θα έχουμε κάποιο είδους λόμπι σε κάθε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε ε, ε, επενδύσεις που να ωφελήσουν τον πολιτισμό. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Η Πρόεδρος, εγώ ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και όλα αυτά συντεριάζουν με την εμπειρία που έχουμε ήδη αποκομίσει. αναφέρατε την Νάντι. Και πήγα εκεί και πήγα με, με το παιδί μου Εκεί μέχρι την παραλία, μέχρι τη θάλασσα δεν υπήρχε τίποτα. Σηκώθηκα και έφυγα. Και ξέρω την αδελφοποιημένη με το Σαρμπρίκεν, την πόλη τη δική μου. Και διαπίστωσα το πώ προχώρησε, πώ αναπτύχθηκε. Είναι καταπληκτικό και τώρα είναι μια όμορφη πόλη. Και το Άρχου επίση επισκεφτήκαμε με κάποια αποστολή. Το φω, το φω, περισσότερο φω. Και ε, κατά κάποιο τρόπο μοιάζει, γιατί είδαμε ότι σε μια σειρά από πόλει που δεν μπορούσαν να έχουν ε, έτσι, ε, ρόδινο μέλλον από, από άλλους τομείς είδαμε πως αναβαπτίστηκαν. Σας ευχαριστούμε και θα πρέπει να υπάρξει το απολογιστικό αποτέλεσμα για να ωφελήσει τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τη μορφή της παρουσίασης πραγματικά έχω να πω μόνο καλά λόγια. Μιλήσατε για την καινοτομία και βεβαίως εδώ υπάρχει μια πολιτική, αν θέλετε, βούληση. Πώς δηλαδή να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, αυτά τα κονδύλια για να προωθήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργικά, καινοτόμα, της σύγχρονης οικονομίας. Τα διαρθρωτικά ταμεία λοιπόν και η στρατηγική του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πολιτιστικά προγράμματα, πολιτιστικούς στόχους. Ο πολιτισμός σαφώς και πρέπει να βρίσκεται σε πολύ σημαντική θέση. Πολιτισμός και πολυμορφία. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να μπορούν να στηριχθούν, να ενισχυθούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί επιτόπου, σε τοπικό επίπεδο, μία ταυτότητα και εγώ γνωρίζω το παράδειγμα κάποιων προγραμμάτων που έχουν πάει πάρα πολύ καλά και στην Εστονία και αλλού στην Ευρώπη και ξέρω επίσης ότι τα θετικά αποτελέσματα πάντα θα πρέπει να στηρίζονται. Βεβαίως εδώ πάντα έχουμε το θέμα του προϋπολογισμού που μας περιορίζει, που μας ε, σταματάει. Είπατε και κάτι πολύ σημαντικό Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, οι οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την εντύπωση και την ιδέα που έχουν ε, οι πολίτες, που αρχίζουν να έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή για βιώσιμη ανάπτυξη, για υφόρο ανάπτυξη. Και αυτό θα πρέπει καταρχήν να το βάλουμε στο μυαλό κάποιων συναδέλφων που ακόμα ανθίστανται. Ευχαριστώ. Σας είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά που μας παρουσιάσατε και εμείς καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός είναι κάτι που έχει πραγματικά λάβει σημαντικές διαστάσεις και στη Γερμανία και αλλού βλέπουμε ότι κάθε φορά που μιλάμε όμως για εξοικονομήσεις το πρώτο που περικόπτουμε είναι πολιτιστικά προγράμματα, είναι ο πολιτισμός. Και αυτό πραγματικά γίνεται και σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και δήμων. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντισταθούμε και όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα έχουμε κάποιες δυνατότητες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Πολλές φορές, όταν μιλάμε για χρηματοδότηση κάποιων ε, καινοτόμων προγραμμάτων, ποτέ δεν σκεφτόμαστε τα διορθωτικά ταμεία όταν πρόκειται για τον πολιτισμό. Και πραγματικά ξέρω ότι στην Περιφερειακή Επιτροπή υπήρχαν κάποιες τροπολογίες που είχαν σαν σκοπό να περιοριστεί το εύρος αυτής της χρηματοδότησης μόνο στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει πραγματικά να χρηματοδοτηθούν και υποδομές. Δεν πρέπει απλώς να περιοριστούμε δηλαδή στο παρελθόν και στη μνήμη, αλλά να δώσουμε και προοπτική στο μέλλον, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική ανάπτυξη. Μας δώσατε πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα και αυτό ήταν κάτι το πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να ενισχύσουμε και αυτό να συνεχίσουμε. Ποια είναι η θετική επίπτωση αυτών των ε, προσπαθειών. Πρόκειται για απτά αποτελέσματα, οικονομικά αποτελέσματα που τα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκο. <clears throat> Ευχαριστώ. Μπράβο κυρία Μοντάλτο. Η μελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί να μας εμπνεύσει στις μελλοντικέ μας δράσεις. Μία ερώτηση. Θέλω να καταλάβω αν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης σας συνειδητοποίησατε τη δυσκολία που έχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες να βάλουν το χέρι πάνω σε αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια γραφειοκρατία που πολλέ φορέ είναι πολύ δύσκολο μερικέ πόλει ή κάποιε περιοχέ, κάποιε περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν του τους αυτού. αυτούς, να έχουν πρόσβαση στους πόρους αυτούς. Βέβαια, από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή ε, αποκτήσουν πρόσβαση, μερικέ φορέ δεν ε, τα ξοδεύουν σωστά. Χθε, συζητούσα με την κυρία Κώστα και ενημερωθήκαμε ότι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν πέρασαν οι τροπολογίες που είχαν σαν σκοπό να προστατεύσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το ότι δεν πέρασαν αυτές οι τροπολογίες στην Περιφερειακή Επιτροπή. Γιατί πρέπει να τονίσουμε αυτή τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το μάθαμε, μας ήρθε ως είδηση. Ελπίζω ότι οι τροπολογίε τουλάχιστον για το νορίζοντα, για το horizon, θα περάσουν. Ευχαριστώ. Να απαντήσω αγγλικά ή ιταλικά. Oh, sorry. Mrs. Costa. κυρία Κώστα, ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη, κυρία Μοντάλτο. Νομίζω ότι φτάνει την κατάλληλη στιγμή, μια επίκαιρη στιγμή, γιατί πραγματικά είμαστε σε φάση όπου ξεκινάει ο προγραμματισμός της νέας εφταετίας. Γι' αυτό λοιπόν και η πρότασή σας είναι πολύ επίκαιρη. Θέλω να πω στους συναδέλφους της ε, Επιτροπής, και ούτως ή άλλως θα το πω και στην έκθεσή μου όταν την ετοιμάσω, αλλά προέκυψε και από τις συζητήσεις της Επιτροπής μας, είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν όντως υπάρχει ένας προσανατολισμός ο οποίος ε, βασίζεται στην αλλαγή του μοντέλου που αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε, να πλασάρουμε, να πουλήσουμε, αν θέλετε, τις ε, πόλεις μας, τις ε, περιφέρειές μας, να δείξουμε τι το ελκυστικό έχουν πολιτιστικά κτλ. Ε, στο πρόγραμμα Regi υπάρχει κάτι τέτοιο. Το λέει αυτό και η, μελέτη σας. Το... Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι το νέο πρόγραμμα και για την ε, καινοτομία και για την ε, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα του πολιτισμού, ε, μειώνεται η στήριξη, η οικονομική στήριξη. Ισχύει αυτό. Εμείς λέμε στην Κομισιόν ότι θα πρέπει να προωθήσει κάποιες οριζόντιες πολιτικές. Όπως λέει και η μελέτη, πρέπει να καταλάβει η Επιτροπή ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένας τομέας, είναι ένας πόρος για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ακριβώς και το περιβάλλον. Πρέπει να το καταλάβει αυτό η Επιτροπή. Αυτή είναι η λογική. Και στη συνθήκη λέγεται ότι ο πολιτισμό είναι οριζόντιο πράγμα και μπαίνει σε όλε τι πολιτικέ. Αλλά αυτό δεν προκύπτει από τον προγραμματισμό που κάνουμε για την επόμενη 7 ετία. Ε, αυτό θα πρέπει να το διατρανώσει και η Επιτροπή Ρέτζι, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης, συμφωνώ με τις συστάσεις σας. Αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός δεν είναι στις 11 προτεραιότητες ε, που αναφέρει η νέα πολιτική συνοχή. έχει ξεχαστεί λιγάκι. Καμπανάκι, καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλο, όλα στο, στα 1,8 δις ε, που δίδονται στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Καλό θα ήταν να γίνει μια συγκριτική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις ε, καλύτερες πρακτικές. Να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός, ούτως ώστε να ενταχθεί ο πολιτισμός σε διάφορες πολιτικές. Υπάρχουν στην Ιταλία ε, βιομηχανικές περιοχές που ήταν βιομηχανικές και που χάρη σε αυτή την προώθηση που τους δόθηκε έχουν μετασχηματιστεί. Ε, επίσης θα πρέπει να δώσουμε κίνητρο στα κράτη-μέλη για να επενδύσουν περισσότερο. Σήμερα, σε επίπεδο εθνικό, έχουμε παντού περικοπές για τον πολιτισμό. Αυτή η πολύτιμη μελέτη σα μα δείχνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η τάση. Νομίζω ότι μα ενημερώνει και μα υπευθυνοποιεί αυτή η μελέτη. Σα ευχαριστώ. Κυρία Παλιαδέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολύ κύριε Μοντάλτο για αυτή την συλλογική δουλειά. Πραγματικά ήρθε σε μια στιγμή που ε, μας αποσχολεί πάρα πολύ η αδυναμία της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την, ε, τον πολιτισμό και την αδυναμία των, ε, των μελών της Επιτροπής Πολιτισμού να πείσουν τις άλλες επιτροπές για την ανάγκη χρηματοδότησης ε, πολιτιστικών δράσεων. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, χρήση του όρου Non-Technological Innovation που μας παρουσιάσατε στην μελέτη σας, γιατί πραγματικά το να ταυτιστεί η καινοτομία όχι με την τεχνολογία αλλά και με μη τεχνολογικές δράσεις είναι μια άλλη προσπάθεια που δύσκολα θα την καταλάβαινε η ΙΤΡΕ, το είδα στο European ε, ε, Institute of Technology ε, που είχα την ευθύνη του. Ε, θα ήθελα κάπου να δω, γιατί δεν ξέρω, αυτή είναι η ερώτησή μου, αν υπάρχει ορισμός για το culture. Ε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι συχνά έχουμε παρανοήσει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε βουλευτής η κάθε επιτροπή, ε, η επιτροπή και το Συμβούλιο τον όρο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Last but Marie Therese. Marie Therese, τελευταία αλλά σημαντική. Merci, Madame. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μοντάλτρο για την έκθεσή της Πλήρη μελέτη. Τα διαρθρωτικά ταμεία με απασχολούν πάρα πολύ γιατί εγώ είμαι μέλος και της Επιτροπής Ρέτζι. Και θέλω να σας ε, επιβεβαιώσω ότι ανησυχούμε και στην Επιτροπή Ρέτζι για αυτό το θέμα. Γιατί κάναμε μια έκθεση πρωτοβουλία, εγώ ήμουν η συντάκτρια του χρο... πέρυσι, για το δυναμικό αυτού του καλλιτεχνικού κλάδου. Και συζητήσαμε και για τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των ε, κλάδων. Ψηφίσαμε κάποιες προτάσεις, ούτω ώστε αυτά τα διαφορετικά ταμεία να χρησιμοποιούνται καλύτερα στον τομέα του πολιτισμού. Μην ξεχνάτε ότι έχει και κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο ο πολιτισμός, αλλά και οικονομικό ρόλο. Είναι διτός ο ρόλος του. Και στην έκθεσή μας ακριβώς λέγαμε αυτά που προτείνετε και εσείς, ίδιες συστάσεις ε, αντιμετωπίσαμε και εμείς τις δυσκολίες που διαπιστώνετε και εσείς. Στον τομέα των διαχωτικών ταμείων ψηφίσαμε στην ε, Επιτροπή αρχές Ιουλίου κάποιες τροπολογίες στον κανονισμό, δηλαδή... Αν είχατε κάνει αυτή τη συνεδρίαση πριν, ίσως θα, ήταν όλα, θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί, αλλά οι διαπραγματεύσει δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Κομισιόν δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα επιμείνουμε ούτω ώστε ο πολιτισμό να φαίνεται περισσότερο στον κανονισμό, ούτω ώστε τις μελλοντικέ εταιρικέ συμβάσει που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα μπει ο πολιτισμός τελικά στα, εκεί, θα μπει στα λειτουργικά προγράμματα και εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να κάνουμε λόμπι στι ε, περιοχέ μας ούτω ώστε να μπει ο πολιτισμό σε αυτά τα προγράμματα, τα επιχειρησιακά ή λειτουργικά. Ε, μιλήσαμε για την πολιτιστική κληρονομιά, μιλάμε για υποδομέ, αλλά υπάρχει και η ανάπτυξη, η ελκυστικότητα που έχει ο πολιτισμό. Ε, όταν υπάρχει πολιτιστικό ενδιαφέρον ας πούμε, σε μια περιοχή είναι πολύ πιο ελκυστικέ. Νομίζω ότι πέρυσι Είχατε παρουσιάσει μια μελέτη με νούμερα πολύ ενδιαφέροντα. Τα νούμερα αυτά θα πρέπει να τα επικαιροποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε το κοινωνικό, οικονομικό δυναμικό ανάπτυξης που έχει ο πολιτισμός. Ε, καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε αυτά τα νούμερα για να εντυπωθούν στον κόσμο, ειδικά σε περίοδους κρίσης όπως τώρα. Merci Je pense aussi qu'il faut parler des routes. Πρέπει να μιλήσουμε και για τις πολιτιστικές οδούς, νομίζω. Πριν από δύο χρόνια είχαμε κάνει λόγο για αυτές. Είναι καλό και για τον τουρισμό και για τον πολιτισμό και για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών μας και περιφερειών μας. Αξίζει της προσοχής μας. Η κυρία Μοντάλτο, έχετε το λόγο. For all... Σε ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας και εγώ με τη σειρά μου να προσπαθήσω επομένως να σας καλύψω και να προσπαθήσω να απαντήσω. Όσον αφορά το, το, τα προβλήματα στην προσβασιμότητα, στα ταμεία, τα, τα διοικητικά προβλήματα, τα προβλήματα από τη γραφειοκρατία, η απάντηση είναι ναι. Αυτό προσπαθήσαμε να το λάβουμε υπόψη. Βέβαια δεν ήταν στο επίκεντρο της μελέτης, όμως βέβαια ε, πρόκειτο για κάτι το οποίο ανέκυψε επανειλημμένος από διάφορους εμπλεκομένους, αρχές, ε, του, του, τους ίδιους τους ε, ασχολούμενους με τα πολιτιστικά και επανειλημμένα είπαμε απομένως ότι τα πολιτιστικά θα πρέπει στα λειτουργικά προγράμματα και στα, στις συμβάσεις ε, εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Γιατί άπαξ και είναι προτεραιότητα τότε δίνονται στα πολιτιστικά χρήματα. Και έτσι είναι πιο εύκολο κανείς με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να έχει πρόσβαση στα ταμεία. Άρα έτσι θα πρέπει να έχουμε ε, ε για, την περίοδο του 2020 καλύτερες διαπραγματεύσεις και βέβαια θα πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα να λυθούν και λύνονται πιο εύκολα σε εθνικό επίπεδο. Βασικό αυτό επίση. Εν γέννη. Σε σχέση με το μας είπατε και ιδίω με αυτά που είπε η κυρία Κώστα για το πόσο σημαντικό είναι το να προσπαθήσουμε να ε, συλλάβουμε ω όχι τομέα, όχι κλάδο, αλλά ως πηγή πολιτικών τον πολιτισμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη στην προσπάθειά μας που γίνεται για να δοθεί ένας ορισμός που είναι τόσο δύσκολο να δοθεί. Όμως το είπαμε και είπαμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να δώσει κανείς ορισμό των πολιτιστικών. Μπορεί κανείς να έχει πρώτα-πρώτα μια φιλοσοφική προσέγγιση. Δηλαδή, έτσι να αντιληφθούμε ως πηγή να συλλάβουμε τα πολιτιστικά και επίσης υπάρχει και ορισμός ε, επί τη βάση των τομέων των κλάδων της οικονομίας ε, υπάρχει ολόκληρη προβληματική προτείναμε εμείς έναν ορισμό που φυσικά επιδέχεται μεταβολές αλλαγές από μια χώρα στην άλλη όμως έτσι να, την, την αντιληφθούμε ως πηγή ανάπτυξης ε, το, τον πολιτισμό και αυτό είναι μια καλή αρχή για να προχωρήσουμε στην απόκτηση κάποιου ορισμού τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη δουλειά μα. Το λάβουμε υπόψη και στην προβληματική για τα διορθωτικά ταμεία. Όχι, δεν είναι αργά. Όλα αυτά τα, τα είχαμε υπόψη μα, αλλά τα δώσατε σε κάποια μορφή, θα συζητήσουμε και σα ευχαριστούμε πολύ χρήσιμα. Και πάλι και πάλι ευχαριστούμε. Σα αξίζουν χειροκροτήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα διάφορα Έχετε να πείτε κάτι για τα πρακτικά. Όχι. Ωραία. 8 και 9 Νοεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση. Μπορείτε να υποβάλλετε και τροπολογίες το συντομότερο δυνατόν στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ τους Γερμηνείς. Και τώρα θα ακολουθήσει και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση των συντονιστών.